Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten... Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε πλούσια ημερήσια διάταξη. Και για να μην ε, καθυστερήσουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα αμέσω. Να περάσουμε με το σημείο 1, έγκριση της ημερήσια διάταξης. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, συμπληρώσεις, παρατηρήσεις. Όχι. Ωραία. Α, παρακαλώ. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Μας ακούτε τώρα. Η Ιταλική διερμηνία υπήρχε πρόβλημα. Εντάξει, όλα είναι εντάξει με τη διερμηνία. Ωραία. Ωραία. Έγκριση λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις, συμπληρώσεις, επιθυμίες. Όχι, ωραία. Εγκρίνεται όσο έχει. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις ε, της Προέδρου. Σήμερα έχουμε διερμηνία στις εξής ε, γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσέχικα, εστονικά, ουγγαρικά, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμανικά και να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται ζωντανή στο ίντερνετ. Τώρα, σας παρακαλώ να αναφερθούμε στο βραβείο Λούξ ε, ως μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε, οπότε σας παρακαλώ και εσείς να ψηφίσετε αν δεν έχετε ήδη ψηφίσει, αλλά να παρακαλέσετε και τους συναδέλφους σας να τους το ξαναπείτε ε, ε, έτσι φιλικά ότι και εκείνοι πρέπει να ψηφίσουν. Νομίζω ότι και τα τρία φιλμ είναι πολύ καλά. Αν δεν τα έχετε δει, να τα δείτε. Αύριο το πρωί, ε, συγγνώμη, σήμερα το πρωί είχαμε μια συνάντηση με την Κομισιόν για το μέλλον αυτού του βραβείου. Δεν προχωρήσαμε πολύ. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο με την κυρία Γκάμπριελ και θα ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά και ελπίζουμε το Δεκέμβριο να προκύψει μια λύση για το μέλλον του βραβείου Λουξ. Αυτές είναι ανακοινώσεις μου. Όπως βλέπετε, ε, το, χώρος ε, είναι λίγο περίεργος και είμαι στο ίδιο επίπεδο με τους συναδέλφους, οπότε είναι ίσως λίγο δύσκολο να δω ποιο ζητάει το λόγο. Σας παρακαλώ λοιπόν να ε, είστε βέβαιοι ότι σας έχουμε σημειώσει εάν θέλετε να πάρετε το λόγο. Δεν υπάρχει καμία κακή πρόθεση, αλλά σε αυτό το δωμάτιο είναι λίγο δύσκολο να σας δούμε καμιά φορά. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσια διάταξης, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που σήμερα για πρώτη φορά Έχουμε τον Επίτροπο Μοσκοβισή εδώ στην Επιτροπή μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήρθε για να συζητήσει με την Επιτροπή μας την σημαντική νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πολιτιστικών θησαυρών. Όπως ξέρετε είναι απαραίτητο να σταματήσει αυτό το λαθρεμπόριο. Και αυτό όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες μορφές ε, εγκληματικότητας, αλλά για να διατηρήσουμε την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται ε, να εισαχθούν στην Ένωση προϊόντα από το Ιράκ και τη Συρία, αλλά δεν υπάρχει κανένα γενικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών θησαυρών. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα αναγκαία, ούτω ώστε η εισαγωγή πολιτιστικών θησαυρών να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο στα, εσωτερικά, στα εξωτερικά σύνορα της ε, Ένωσης. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, του χρόνου δηλαδή, πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία ακριβώς της πολιτιστικής κληρονομιάς Σημαντική λοιπόν είναι η πρωτοβουλία της Κομισιόν, είναι ένα συγκεκριμένο μέτρο για να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ε, κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, όχι μόνο την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Και γι' αυτό φυσικά την χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα θα ακούσουμε τι περιέχει αυτή η νέα πρόταση στην ε, επεξεργασία της, από ό,τι φαίνεται, θα συμμετάσχουμε με βάση το άρθρο 54 του εσωτερικού κανονισμού. Κύριε Επίτροπε, να ακούσουμε την παρουσίασή σας και φυσικά αν θέλετε να αναφερθείτε και σε άλλα θέματα, έχετε κάθε δυνατότητα, έχετε το λόγο για περίπου 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, και κύριοι Αντιπρόεδροι, αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Δεν έχω ακόμα την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτή την Επιτροπή, παρότι είχα διμερείς επαφές με κάποιους από εσάς σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση και μεγάλη μου τιμή επίσης να βρίσκομαι μεταξύ σας σήμερα. Μπορεί να φανεί περίεργο. Είμαι επίτροπος μακροοικονομικών θεμάτων, οικονομικών, φορολογίας και θα αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο να έρθω στην Επιτροπή Πολιτισμού. Πώς σχετίζονται τα θέματα της φορολογίας με τις εργασίες σας. Και όμως επηρεάζουν πολύ σημαντικά τον κόσμο του πολιτισμού ε, και μάλιστα αφορούν και την επικαιρότητα. Την επικαιρότητα ε, που αφορά τους πλούσιους, τη φορολογία. Εδώ και τρία χρόνια προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή ε, από το γραφείο μου του Επιτρόπου. Είναι σημαντικά θέματα και μερικές φορές δύσκολα για τους συμπολίτε μας με τα Paradise Papers. Σκοπός είναι να καταπολεμήσουμε επίσης και τη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Έτσι λοιπόν τα πολιτιστικά αγαθά είναι ένας από τους ε, πόρους ε, χρηματοδότησης τέτοιου είδους. Γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα. Η Παλμύρα, η Νιμρούντ, η Νινεβή είναι γνωστά σας ονόματα. Διότι όλες αυτές οι τοποθεσίες ε, τις έχουμε δει στις ειδήσει τους τελευταίους μήνες, έχουμε δει τις τραγικές τρομακτικές εικόνες ε, αρχαιολογικών χωρών που καταστράφηκαν από το Ισλαμικό κράτος. Αρχαιολογικοί χώροι ανεκτήμητης αξίας ε, ε, διαγράφηκαν από το χάρτη. Αυτές οι καταστροφές μας διηγούνται όμως μόνο μία, ένα κομμάτι της ιστορίας. Ορισμένα από τα αρχαία που λαιλατήθηκαν από αυτούς τους χώρους πουλήθηκαν ξανά στην Μέση Ανατολή ή στις ευρωπαϊκές αγορές. Πέραν λοιπόν των θεατρικών αυτών καταστροφών ε, που διέπραξε το Ισλαμικό κράτος για λόγους προπαγάνδας και ιδεολογίας έχουμε ε, και άλλα κίνητρα, πολύ πιο πραγματικά, πιο ρεαλιστικά, οικονομικά κίνητρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια τεράστια διακίνηση έργων τέχνης διακίνηση η οποία χρηματοδοτεί με τη σειρά της τις τρομοκρατικές ενέργειες του Ισλαμικού κράτους. Αποτελεί πηγή εσόδων ε, όπως η λελεσία τραπεζών, όπως οι φόροι που επιβάλλονται σε τοπικούς πληθυσμούς, όπως ο έλεγχος των πετρελαϊκών πηγών. Ε, αυτή τη στιγμή, ναι, κερδίζουμε φυσικά τη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους, αλλά οι τρομοκράτες, όπως βλέπουμε, κάθε εβδομάδα εξακολουθούν να είναι ζωντανοί. Είναι διπλό λοιπόν το διακύβευμα, αφενός πολιτιστικό που ενδιαφέρει εσά θέμα ασφαλείας φυσικά ε, και οικονομικό. Η Επιτροπή γνωρίζει απόλυτα ε, πόσο τεράστια είναι αυτή η πρόκληση του παράνομου εμπορίου ε, πολιτιστικών αγαθών. Πέρα από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα έσοδα συμβάλλουν και στη οργανωμένο έγκλημα, στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε κάτι που μας απασχολεί εμάς συγκεκριμένα την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Πέρυσι ε, το τελωνείο οι τελωνιακές υπηρεσίε στο αεροδρόμιο Ρουασί ε, στη Γαλλία κατέσχεσε ανάγλυφα που προέρχονταν από την, περιοχή, ε, από την εμπόλεμη περιοχή της Συρίας και του Ιράκ. Τα, είχαν προσπαθήσει να τα εισάγουν ως διακοσμήσεις κήπου, ως διακοσμητικά κήπου και ο τρόπος με τον οποίο είχαν συσκευαστεί ανακοίνησε τις υποψίες των, τελωνιακών, των καλών τελωνιακών και άνοιξαν τα πακέτα για να δουν από πού προέρχονταν αυτά τα ανάγλυφα. Και αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Τρανταχτή επιτυχία δυστυχώ σπάνια. Σπάνια γιατί, διότι έτσι όπω έχουν τα πράγματα σήμερα, είναι δύσκολο να καταπολεμήσουμε τόσο αποτελεσματικό όσο θα θέλαμε ε, αυτό το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών. Γιατί, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό πλαίσιο για το θέμα αυτό, μόνο εθνικές νομοθεσίες οι οποίες πολλές φορές διαφέρουν, όχι πάντα αποτελεσματικές ε, και όχι πάντα ισότιμες και οι εγκληματίες, οι τρομοκράτες είναι οι πρώτοι που εκμεταλλεύονται αυτά τα κενά. Γι' αυτό τον λόγο, πέρυσι τον Ιούλιο, η Κομισιόν υιοθέτησε μια πρόταση κανονισμού που επιβάλλει τελωνιακού ελέγχου ε, στι εισαγωγέ πολιτιστικών αγαθών, ε, αυτών που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Η πρόταση είναι ουσιαστικά επιχειρεί να αποτελέσει τροχοπέδι σε αυτή τη διακίνηση, απαγορεύοντα την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πολιτικών αγαθών που έχουν εξαχθεί παράνομα από τι χώρε καταγωγή του. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση παρέχει στι τελωνικέ αρχέ τα μέσα να ε, ανακόψουν αυτή την εμπορία πολιτιστικών αγαθών. Αυτό βασίζεται πάνω σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό ορισμό των εισαγόμενων πολιτιστικών αγαθών, καλύπτει μεγάλη ποικιλία αντικειμένων, αρχαιολογικών αντικειμένων, ε, παλιών εγγράφων, ε, έργων τέχνης, ε, ιστορικών. Δεύτερον, θέλουμε να καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τα έγγραφα. Πρέπει δηλαδή όποιο κάνει εισαγωγέ να έχει ειδικέ άδειε εισαγωγή για τα αγαθά αυτά, αρχαιολογικά είδη, χειρόγραφα, και για τα άλλα πολιτιστικά είδη οι εισαγωγή θα πρέπει να ε, υποβληθούν σε ένα σύστημα πιστοποίησης πιο αυστηρό που θα πιστοποιεί ότι η εξαγωγή έγινε νόμιμα. Ουσιαστικά μιλάμε για εχνηλασιμότητα των πολιτιστικών αγαθών τρίτων για την υλοποίηση. Οι τελικέ αρχέ θα μπορούν να κατασχέσουν και να διατηρήσουν τα αγαθά όταν δεν έχει αποδειχθεί ότι εξήχθησαν ε, νόμιμα. Θέλουμε λοιπόν να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες των τελωνίων στα ε, αγαθά τα οποία δεν τρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Γι' αυτό θα ε, επικεντρωθούν στα αγαθά ηλικίας άνω των 250 ετών. δεν είναι φυσικά ο ορισμός, ο κλασικός ορισμός των αρχαίων, αλλά αυτό θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στα, πιο ε, στα αγαθά που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο και δεν θα περιορίσουμε έτσι τη διακίνηση ε, σύγχρονων έργων τέχνης ε, και θα βοηθήσουμε να γίνουν πιο αποτελεσματικέ στου ελέγχου του οι τελωνικέ αρχέ. Γι' αυτό το λόγο αυτή η νομοθετική πρόταση θα ενισχυθεί με μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση για τους πιθανού αγοραστέ και ανάθεση ευθυνών θα έλεγα στους αγοραστές αυτούς ε, μέσω της ε, κατάρτισης των τελωνιακών σε συνεργασία με την UNESCO. Ε, η πρόταση αυτή αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου της Κομισιόν κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Δεν θα επεκτάθω σε αυτό. Μου ζητήσετε να είμαι σύντομο. Έχουμε επικαιροποίησει τους κανόνες ελέγχου ε, εισόδου και εξόδου μετρητών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας το έχουν ζητήσει ε, γιατί αυτά τα χρήματα χρηματοδοτούν τα τρομοκρατικά και τα εγκληματικά δίκτυα. Είχαμε μια πρόταση από τον Δεκέμβριο του 2016 που αυτή τη στιγμή συζητείται στο κοινοβούλιο σας στο δημοσιονομικό, στο φορολογικό τομέα. Ασχολούμαστε με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που χρησιμοποιείται επίσης για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Η απάτη ε, διασυνοριακού ε, ΦΠΑ εκτιμάται στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οπότε πέρυσι προτείναμε πλήρη ε, αναδιάρθρωση του συστήματος του ΦΠΑ ώστε αυτές οι διασυνοριακές συναλλαγές να αντιμετωπίζονται ως εθνικές ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα 40 από τα 50 δισεκατομμύρια που αναφέρα. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αφορά επίσης και το Κοινοβούλιο ε, και έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τους συναδέλφους σας ε, για το θέμα αυτό. Με τα σκάνδαλα που όλο ένα εμφανίζονται, έχουμε τα Paradise Papers αυτή τη στιγμή, ε, όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι να συμβάλλει ο καθένας δικαίως στο φορολογικό σύστημα αυτό αποτελεί το επίκεντρο των δημοκρατικών διαδικασιών ε, αναμφίβολα σε ένα κράτος, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον συνονούν όλοι ε, οι πολίτες ε, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί κατάλληλα. Και αυτό θα γίνει και με ένα θέμα που είναι προσφυλές στη Δική Επιτροπή, την εκπαίδευση, την παιδεία των νέων. Θα κλείσω ε, για να σα αναφέρω αυτό που ξεκινήσαμε χθε, την εκστρατεία που ξεκινήσαμε χθε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ευαισθητοποιήσουμε του νέου μέσω και τη UNESCO, μέσω αλληλεπιδραστικών σελίδων στο διαδίκτυο, μπορούν να καταλάβουν οι νέοι πώ χρηματοδοτούνται οι δημόσιε υπηρεσίε του ε, τα γήπεδα αποδοσφαίρου τα σχολεία τους και όλα αυτά και έτσι θα καταλάβουν γιατί μία μέρα θα κληθούν ως Ευρωπαίοι πολίτες να πληρώνουν φόρους. Αυτά ε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είχα να πω σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση να σας πω ότι υπολογίζω φυσικά στην Επιτροπή σας ε, ώστε να έχουμε μια γρήγορη έγκριση αυτής της πρότασης που πιστεύω είναι γενικού ε, συμφέροντος, ε, γενικού ενδιαφέροντος, κοινού ενδιαφέροντος αφορά οικονομικά θέματα, θέματα ασφαλείας, πολιτιστικά θέματα, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. μην ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό πράγματι αυτό το θέμα του πολιτισμού. Το θέμα αυτό του πολιτισμού θα αναφερθεί στο Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου. Ε, πολλά κράτη-μέλη ξέρω ότι θέλουν να κινηθούμε γρήγορα και χαίρομαι γι' αυτό. Όλα αυτά αποτελούν κομμάτι ενός σχεδίου δράσης ε, πολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατία που υιοθετήθηκε ήδη πριν από ένα χρόνο. Οπότε είναι πολύ φυσικό να υπάρχει αυτός ο χαρακτήρα κατεπήγοντο ε, σε αυτή τη μάχη, την οποία ναι, κερδίζουμε όλο και περισσότερο, αλλά που σίγουρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις. ganz, ganz Dank. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτροπέ για την παρουσίασή σας και την πολύ σημαντική θεωρώ πρωτοβουλία σας και θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και ιδίω η Επιτροπή μας οπωσδήποτε ενδιαφέρεται να προχωρήσει ταχαίως το θέμα αυτό γιατί επίκειται και το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς ε, το επόμενο, θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα λοιπόν ότι δεν ενδιαφερόμεθα μόνο για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και δεν λέμε μόνο λόγια, αλλά είμαστε διατεθειμένοι και σε θέση να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να διασώσουμε και να προστατεύσουμε και τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια πολιτιστικά αγαθά. Να δώσω πρώτα το λόγο στους συντονιστές εφόσον ε, το επιθυμούν και κατόπιν και στα ε, υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Λοιπόν, για το ΕΛΚΑ είναι ο κύριος Στογεύσκη. Παρακαλώ, δύο-τρία λεπτά κύριε Στογεύσκη. Για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε, έχω τρεις ερωτήσεις. Εν είδη συντόμου εισαγωγής να λάβετε υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο έργων τέχνης επί πολλά έτη λαμβάνει η χώρα όσο θεωρούμε ε, πολύτιμα και ακριβά τα έργα τέχνης. Ε, όσο υπάρχει αυτή η αντίληψη υπάρχει αυτό το εμπόριο. Στην Ευρώπη ε, έχουμε βελτιωθεί όσον αφορά την ανακάλυψη του παρανόμου, του λαθρεμπορίου έργων τέχνης. Έχουμε, παραδείγματος χάρη μας ενημερώνουν και οι οίκοι δημοπρασιών δεν είμαστε τόσο καλοί όσον αφορά την ε, πώληση αυτών των έργων τέχνης στο διαδίκτυο, online. Ερώτηση. Ε, έχει διαρευνηθεί το θέμα αυτό το εμπορίου έργων τέχνης στο διαδίκτυο. Μετά, ήμουν υπουργό πολιτισμού για μία επταετία κατά το παρελθόν και ήμουν πολύ δραστήριο όσον αφορά την επιστροφή κλαπέντων ε, αντικειμένων τέχνης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος, πρέπει να το πω, στην Ευρώπη. Όσον αφορά τη συνεργασία όμως με τη Ρωσία, εδώ η κατάσταση είναι αρκετά σκοτεινή. Κάνετε κάτι σε αυτό το τομέα όσον αφορά τη Ρωσία. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση. Τρίτη ερώτηση. Τουρκία. Ο μεγαλύτερος αριθμός έργων τέχνης από το Αφγανιστάν, τη Συρία και από άλλες χώρες ήρθε στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας και δόθηκαν διάφορες πληροφορίες περίπου 4.000 αντικείμενα μέχρι, ένα, μέχρι εκατομμύρια αντικείμενα 400.000 μέχρι εκατομμύρια αντικείμενα ξέρετε τίποτα περισσότερο πάνω σε αυτό Ευχαριστώ πολύ Σίλβια Κώστα για τους σοσιαλιστές Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πολύ σημαντικό να είσαστε εδώ παρόν σήμερα. Θα ήθελα να πω εν γέννη ότι δεν με εκπλήσει καθόλου που ο υπεύθυνο για το θέμα αυτό που αφορά φυσικά την οικονομία και τη φορολογία και τα δημοσιονομικά πέρα από τα τελωνία να ασχολείται και με τον πολιτισμό. Διότι πιστεύω ότι ο πολιτισμός είναι ένας από τους άξονες ανάπτυξης και παραγωγής πλούτου και ίσως από αυτή την πτυχή θα ήθελα να δεσμευτείτε ε, ούτω ώστε να έχει προτεραιότητα στην Επιτροπή Γιούνκερ η ε, λέξη πολιτισμό. Σήμερα δεν αναφέρεται. Όσον αφορά αυτή τη σημαντική οδηγία, ήδη μετά, μετά την καταστροφή της Παλμύρας, σαν Επιτροπή Πολιτισμού σε επίπεδο UNESCO Europol, είχαμε διοργανώσει συναντήσεις και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ζητήσαμε να θεωρηθεί ε, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας η καταστροφή του πολιτιστικού ε, πολιτισμού και ζητήσαμε αυτή την οδηγία που ακόμα δεν υπήρχε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που προτείνεται τώρα. Ε, να επισημάνω κάτι όσον αφορά την οδηγία, δηλαδή ότι αναφέρεται μονάχα στους ελέγχους από το ελληνικές αρχές. Σε πολλές χώρες, όπως και στη δική μου, είναι αναπτυγμένη πολύ σημαντική δράση από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα μπορούσε αυτό να γίνει κοινή προσπάθεια με τους άλλους φορείς. Θεωρώ που ανέφερε ο συνάδελφος, ο προλαλής σας, να μην εξετάσουμε μόνο τη φυσική εξεταστατελωνία, τα φυσικά αντικείμενα, αλλά τι γίνεται και στο διαδίκτυο, online, το εμπόριο, το ελευθερεμπόριο online. Χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Μετά η φορολόγηση δεν μας ενδιαφέρει μόνο το σημαντικό το θέμα της πρόληψης της φοροδιαφυγής που συμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά να προσέξετε επίσης τη φοροδιαφυγή των over the top όσον αφορά τα πολιτιστικά αυτά ε, αντικείμενα. Δηλαδή, θε, μειωμένη φορολογία όσον αφορά το ΦΠΑ για τα πολιτιστικά προϊόντα κυρίως τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα e-books. Ε, νομίζω ότι συζητείται και στο Συμβούλιο αυτό. Μετά, είναι σημαντικό ε, αυτό που είπατε στο τέλος, καλύτερη προστασία και επίγνωση από πλευράς των πολιτών και της νέας γενιάς της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει επένδυση στην κατάρτιση, στην παιδεία όσον αφορά την κληρονομιά αυτή. Ξεκινώ στην αφετηρία. Το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το φως και της όλης προβληματικής που αφορά και το διαπολιτισμικό διάλογο, την όλη αντίληψη της πολιτιστικής κληρονομιάς που θα είναι αντικείμενο του χρόνου συγκεκριμένης χρονιάς και του πολιτισμού σαν νέας άξονας ανάπτυξης πώς, τι θα κάνετε να μπει στο επίκεντρο και μακροοικονομικά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο τομέας του πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χουντής από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μοσχοβησή, σας καλωσορίζω στην Επιτροπή. Ήταν ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας κάνετε των πρωτοβουλειών που εν γέννη παίρνει η Κομισιόν με την ευκαιρία του 2018 έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και για την παρουσίαση του συγκεκριμένου κανονισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι εδώ είναι ο αρμόδιος επίτροπος, θέλω να θυμίσω μια αντίστοιχη σημερινή λαιλασία δημόσιας περιουσίας και δημόσιων αγαθών που γίνεται στην Ελλάδα. Τα ελληνικά αεροδρόμια τα έχουν πάρει οι Γερμανοί, τα ελληνικά, τους ελληνικούς συνδροδρόμους οι Ιταλοί, το νερό στους Γάλλους και τα υπερκέρδη των, των ελληνικών ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα λέω αυτά για να πάρει ο κύριος Επίτροπος τις αντιστοιχίες. Στον τομέα του πολιτισμού, κύριε Επίτροπε, έχει επέλθει μια λαιλασία που κρατάει χρόνια έτσι, λασία έργων τέχνης και αρχαιότητας στην Ελλάδα, έτσι. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα τα έχουν οι Βρετανοί. Τα αγάλματα της νίκης της Αμμοθράκης και της Αφροδίτης της Μήλου στο Λούβρο στη Γαλλία. Αρχαιότητες και έργα τέχνης εκλάψαν και απομακρύνθηκαν από την Ελλάδα λόγω της ναζιστικής κατοχής. Σας ερωτώ λοιπόν κύριε Επίτροπε, ως Έλληνας Ευρωβουλευτής, αλλά και ως εισηγητή στην γνωμοδότηση που με έκανε την τιμή η Επιτροπή για την ε, οδηγία που μιλάμε για τι συνοριακές αιτήσει επιστροφής έργων τέχνη που λαιλατήθηκαν σε περίοδο ένοπλων συγκρούσεων. Θα ήθελα λοιπόν, επαναλαμβάνω, να σα ρωτήσω, θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία σχετικά με αυτά τα, τις και τις ε, έργα τέχνης που έχουν φύγει από τις χώρες προέλευσης, τις χώρες παραγωγής ε, και αναφέρονται στα συγκεκριμένα αυτά θέματα. Διότι διαφορετικά, επιτρέψτε μου και τελειώνω με αυτό κύριε Επίτροπε, αυτά που λέτε εσείς, αυτά που θα πούμε και εμείς, περί ευαισθησίας, περί προστασίας της κοινή πολιτιστικής μας κληρονομιάς και περί έτους σε αυτά, ακούγεται πολύ υποκριτικά και δεν πείθει για την αγαθότητα των προθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο η Χέλγα για τους πρασίνους. Ευχαριστώ Πέτρα. Είναι πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα. Και μας αφορά πραγματικά. Είναι τρομακτικό αυτό που κάνουν οι τρομοκράτες. Τα ανθρώπινα όντα έχουν την ικανότητα να καταστρέψουν τον πολιτισμό και ανθρώπους ε, για ιδεολογικού λόγου. Και είναι τόσο δύσκολο να του πολεμήσει κανεί γιατί αισθάνονται ότι έχουν μια αποστολή, ότι έχουν το δικαίωμα να καταστρέψουν πολιτιστικά αγαθά και έργα διότι θεωρούν ότι δεν είναι... ανταποκρίνονται στι θρησκευτικέ του πεπιθήσει ή οτιδήποτε. Ε, πιστεύω λοιπόν ε, αυτή τους υπεποίθηση ότι είναι ήρωε ήρωες καταστρέφοντας ε, το δυτικό πολιτισμό ή τον ελληνικό πολιτισμό αλλά όχι το δικό τους γι' αυτό το, γι αυτό το λόγο είναι τόσο δύσκολη η καταπολέμηση του. διότι ελάχιστε είναι οι δυνατότητε που έχουμε. Ή δεν μπορούμε να του πείσουμε, το οποίο όπω φαίνεται είναι αδύνατο, ή να του πολεμήσουμε, το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ή μπορούμε επίση να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα χρήματα που κερδίζουν πουλώντα αυτά τα παράνομα ε, έργα τέχνης. Ε, και αυτή είναι η μπορουμε επιση να προσπαθησουμε να περιορισουμε τα χρηματα που κερδιζουν πουλωντα αυτα τα παρανομα εργατεχνη και αυτη ειναι η ερωτηση προ εσά, κύριε Μοσκοβισή. Τι γίνεται με ε, τις πετρελαϊκές ε, δραστηριότητες ε, με τις οποίες χρηματοδοτούν τις δικές τους τρομοκρατικές δραστηριότητες. Πώς θα περικόψουμε αυτούς τους πόρους που τους ενδυναμώνουν. Δεν είναι μόνο το παράνομο εμπόριο, δηλαδή έργων Αυτό πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε είναι και τους άλλους οικονομικούς πόρους της Αλκάιντα και όλων των υπολείπων τρομοκρατικών οργανώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πίτροπε, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Πολλά υπόθηκαν, δεν θα πω πολλά. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσετε στην ερώτηση της Χέλικα Τρίπελ σε πέντε λεπτά και συμφωνώ με αυτά που είπε ο στο Υπάρχει διεθνής διάσταση. Υπάρχει. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία και τη Ρωσία. Και στη Συρία και τη Λιβύη δεν ξέρω τώρα βέβαια με ποιους θα συνεργαστούμε. Και το βαθύ ίντερνετ επίσης. Εκεί ε, διεξάγεται πολύ εμπόριο. Προσπαθούμε βέβαια να ε, το ελέγξουμε, αλλά δεν νομίζω ότι επιτυγχάνουμε σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε μέχρι πότε θα πρέπει να περιμένουμε για να εγκριθεί αυτός ο κανονισμός. Θα προλάβουμε να τον εγκρίνουμε κατά την τρέχουσα θητεία μας ή θα πάρει πολλά χρόνια ο, η πρόεδρος. Μα έχει να κάνει και με εμά το Κοινοβούλιο, αλλά βέβαια και με το Συμβούλιο. Τώρα, η κυρία Μπίλτα και μετά θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο, αλλά η κυρία Μπίλ θα κλείσει τον ε, πρώτο γύρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε όσον αφορά την πρόταση κανονισμού. Πιστεύω ότι όλοι συνεκλονίσαν από τις εικόνες που είδαμε των τζιχαντιστών που καταστρεφάν πολύ παλιά γάλματα χιλιετιών και μνημεία χρησιμοποιώντας εκρηκτικά χωρίς να σέβονται τίποτα. Πιστεύω τέλος ο κόσμος τα είδε αυτά Λοιπόν, η UNESCO αποκάλεσε γενοκτονία πολιτιστική. Αυτό το γεγονός είναι ισχυρός όρος, θα έλεγα, αλλά νομίζω ότι αυτό δείχνει αυτές τις πράξεις όσον αφορά το παράνομο εμπόριο των πολιτιστικών έργων, ακόμα και αν δεν ειδηγούν στην καταστροφή των έργων αυτών. Επίσης ε, είναι βλάπτη τον πολιτισμό, διότι παίρνει τη φυσική κληρονομιά ενός πολιτισμού ε, και απαλλάσσει, τους παίρνει τη μνήμη τους αν θέλετε και την ιστορία τους. Το Ισλαμικό κράτος και στομοκριτικές ομάδες και τέτοιες πρακτικές για τη χρηματοδότηση των εγκλημάτων τους θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους το εμπόριο. Αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να καταπολεμήσουμε την εκρίζωση των πολιτιστικών αυτών αντικειμένων. Οι αρπάρκειες αυτών των αντικειμένων ε, ε, εμποδίζει εκείνων που κληρονομούν αυτά τα αντικείμενα να αξιολογήσουν τη σημασία που έχουν τα αντικείμενα. Για μία ακόμη φορά, μέσω όλων αυτών των προγραμμάτων, σχεδίων και εξέταση των θεμάτων, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρωταρχικό είναι ότι θα πρέπει να επανέλθουμε να βάζουμε τα σύνορα, διότι είναι ο μόνος τρόπος τα σύνορα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να δώσω το λόγο τώρα πρώτα απ' όλα στον κύριο Μοσκοβισή για να απαντήσει και μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχω Μέσιους, Φλίν, Βόρντ, Σαμιντίμιτς και Κριστίνα Λιμπάτσκα στο δεύτερο αυτό κατάλογο. Λουίτζι Μόργαν επίσης. Και έτσι θα έκλεινα τον ε, κατάλογο μιλητών γιατί αλλιώς θα καθυστερήσουμε. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ οι δυνατόν πέντε λεπτά αν είναι δυνατόν σε πέντε λεπτά. Θα προσπαθήσω. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στη συζητήση σας. Θα ήθελα να μπορούσα να απαντήσω σε όλα. Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα για τα θέματα αυτά, αλλά εδώ είμαι επίτροπος της φορολογίας και των τελωνίων για να ασχοληθούμε με πολύ συγκεκριμένα θέματα. Αλλά φυσικά όλα αυτά που λέτε είναι πραγματικά συναρπαστικά. Πρώτα απ' όλα, Ποια είναι η προσέγγιση μας. Μιλήσατε για πολιτιστική γενοκτονία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο γενοκτονία ε, εύκολα, αλλά είναι σίγουρα λασία, είναι καταστροφή και επιπλέον ε, αξιοποιείται για να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες καταστροφικές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί. Η πρόταση αυτή ασχολείται με την δραστηριότητα των τελωνίων. Δεν είναι μια πρόταση που προσπαθεί να εκαθιδρύσει συνεργασίες. Μόνο ελέγχος. Θέλουμε να ελέγξουμε τις ροές εμπορευμάτων ανεξάρτητα από την προέλευσή τους είτε προέρχονται από ζώνες συγκρούσεων που πρέπει να ελέγχονται φυσικά και ακόμη και αν περνάνε από τρίτες χώρες όπως η Ρωσία και η Τουρκία. Δηλαδή αυτό το οποίο έμεσα ε, πρέπει να εξετάσουμε είναι η ποιότητα της ε, τελωνιακής μας συνεργασίας. Βεβαίως με την Τουρκία έχουμε μια ε, πολύ ανεπτυγμένη συνεργασία. Η πρότασή μας αφορά το διεθνές λαθρεμπόριο και μου ζητήθηκε να απαντήσω εάν τα τελωνία εργάζονται μόνο τους. Όχι εργάζονται στα πλαίσια ενό ε, ευρυτέρου δικτύου, συνεργάζονται με τα Υπουργεία Πολιτισμού, για παράδειγμα. Όταν πρέπει να ζητηθούν πιστοποιητικά. Αυτό γίνεται για να έχουμε αυτή την ανιχνευσιμότητα στην οποία αναφέρθηκα. Ε, μου τέθηκε ένα ερώτημα για τις ε, ηλεκτρονικές δημοσίευσεις. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για τη στήριξή της στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους συντελεστές, για τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα e-book και άλλες δημοσιεύσεις ε, στο ίντερνετ. Είμαι πεπισμένος ότι είμαστε στον 21ο αιώνα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση γενικότερα στις ηλεκτρονικές ε, δημοσιεύσεις, ισότιμη προς τις ε, έντυπες δημοσιεύσεις. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής υπό την Προεδρία της Μάλτας διότι ε, ένα μόνο κράτος μέλος, η τσεχική δημοκρατία, έχει μπλοκάρει το θέμα για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με, με τις δημοσιεύσεις. Ε, ξέρετε πώς γίνεται, αξιοποιούν ένα θέμα για να αποκτήσουν κάτι σε κάποιο άλλο. Και φοβάμαι ότι και κατά την Εστονική Προεδρία δεν θα καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική λύση. Υπάρχουν ε, εκλογές στην Τσεχία. Περιμένω η νέα κυβέρνηση να βοηθήσει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν και στην ουσία συμφωνεί και η Τσεχία. Αλλά θέλει ε, να ξεπεράσει με αυτή τη στάση κάποιο άλλο πρόβλημα, σε κάποιο άλλο θέμα. Τώρα για τον έλεγχο των εισαγωγών των πολιτιστικών αγαθών, βεβαίως είναι σοβαρή ανησυχία μας, γιατί δεν πρέπει να γίνεται αυτό το λαθρεμπόριο και η πρόταση που υιοθετήθηκε τον ε, Ιούλιο θα σταματήσει την παράνομη, το λαθρεμπόριο λοιπόν πολιτιστικών αγαθών που εξάγονται από τις χώρες προέλευσης. Είναι μια πρόταση που αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα, όχι. Όχι, συμμετέχουμε, ε, συμμετέχουν σε την προσπάθεια και άλλοι οργανισμοί, UNESCO, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Οργάνωση Τελωνίων, το G7. Η κυρία Τρίπελ έθιξε ευρύτερα θέματα δεν έχω απάντηση, σημειώνω. Για παράδειγμα, πώς αξιοποιούν το λαθρεμπόριο πετρελαίου, ιδιαίτερα μέσω της Τουρκίας. Θα μπορούσαμε να εξυγχρονίσουμε την ε, τελωνιακή μας συνεργασία με την Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Βεβαίως, η πρότασή μου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αλλά πιστεύω ότι είναι και ζωτική σημασία από μόνη της. Και ελπίζω, αυτό βέβαια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εσά, να εγκριθεί κατά τη διάρκεια τη τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Εγώ θα ήλπιζα να εγκριθεί αρχέ ε, του 2018 για να εφαρμοστεί, γιατί δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Δεν σταματάει ούτε το λαθρεμπόριο ούτε η τρομοκρατία. Πρέπει λοιπόν και εμεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Τώρα για την Ελλάδα φυσικά δεν θα απαντήσω ε, βέβαια τη χώρα σας, την αγαπώ πάρα πολύ και με απασχολεί πολύ. Τώρα εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω εάν τα μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να είναι στην Ακρόπολη στο Βρετανικό Μουσείο. Ξέρω ότι υπάρχει σοβαρή και με παλιά ιστορία σύγκρουση από αυτού. Είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι πρέπει να μας αντιμετωπίσει ευρύτερα, αλλά δεν είναι αντικείμενο της παρούσης προτάσεως. Αλλά βεβαίω όλοι είμαστε ευαίσθητοι απέναντι του θέματος αυτού. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάθιος παρακαλώ. Σας παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση για το νόμιμο εμπόριο ε, έργων τέχνης ε, και αρχαίων αντικειμένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι νέοι μας ε, πολίτες για να εκτιμήσουν σωστά τον πολιτισμό των άλλων χωρών πρέπει να μπορούν να τα δουν από κοντά αυτά τα αντικείμενα, να μπορέσουν να, τα, να έρθουν σε επαφή με αυτά. Οπότε εκτιμάμε ιδιαίτερα τα βήματα που κάνετε για την καταπολέμηση της λαιλασίας τέτοιων ειδών, αλλά δεν θέλω οι προσπάθειες αυτές να παρεμποδίσουν το νόμιμο εμπόριο διότι είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι μιας χώρας να μπορούν να πάνε σε ένα μουσείο ή σε μια συλλογή και να δουν ε, έργα τέχνης, ε, αρχαία είδη από άλλες ε, χώρες. Θέλουμε να κατανοήσουμε, να μάθουμε τις ζωές και τους πολιτισμούς άλλων χωρών. Οπότε το νόμο εμπόριο αρχαίων ειδών και έργων τέχνης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να παρεμποδιστεί κατά κανέναν τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όφλιν. Ευχαριστώ πολύ. Να σας συγχαρώ κύριε Επίτροπε, κύριε Μασχοβησή για ε, το, ενασχόλησή σας με αυτό το ζήτημα του λαθρεμπορίου πολιτιστικών ειδών. Είμαστε στο πλευρό σας και θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας για να σας ρωτήσω δύο ερωτήματα πιο γενικής φύσης. Πρώτον, νομίζω ότι έχω δίκιο λέγοντας ότι αναμένουμε μια πρόταση της Κομισιόν κάποια στιγμή μέσα στο έτος ε, για να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ε, για την κάλυψη του ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών. Ε, αυτό αφορά και το ζήτημα της φορολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, υγειονομικών προϊόντων γυναικείων ε, και, και ο κύριος Μάθιος είχε επιχειρηματολογήσει γι' αυτό. Είχε τεθεί αυτό το θέμα με το Ηνωμένο Βασίλειο. πρόκειται να δούμε μια πρόταση σύντομα. Δεύτερον, η Κομισιόν σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες μας στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο κατά 15% ή τόσο ουσιαστικά είναι η συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα, συμπεριλάβετε, θα συμπεριλάβετε κάποιες πληρωμές αναχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ώστε να απαλύνεται το πλήγμα. Υπάρχει κάποιο σενάριο ήδη ρεαλιστικό και μετά τα προγράμματα δαπάνης ε, σε πολιτιστικούς, ε, στον πολιτιστικό τομέα πρόκειται να μειωθούν ε, ε, μέσα στο... Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τέτοιο. Ε, Ward, Ευχαριστώ, Julie Ward, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να μην μιλήσουμε μόνο για πολιτιστικά αγαθά, αλλά να θυμηθούμε τους καλλιτέχνες και τους ακτιβιστές στον τομέα τον καλλιτεχνικό που έχασαν τη ζωή τους τον Καλέντ Αλαλσάντ που ήταν 81 ετών αρχαιολόγος που πρόσεχε το Μουσείο της Παλμύρας στη Συρία επί 40 χρόνια και δολοφονήθηκε και τον Μπασέλ Κάτεμπιλ εκείνο που είχε αναπτύξει λογισμικό ανοιχτή πηγής και δημιούργησε ανοικοδόμηση της διάστατη εικονική της αρχαίας πόλης και είπε η χείρα του ότι σκοτώθηκε τον Αύγουστο, πέθανε τον Αύγουστο αλλά ανακάλυψαν ότι είχε πεθάνει δύο χρόνια πριν. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι σε αυτή τη φιχτή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, Σύριοι και Μουσουλμάνοι είναι τα θύματα κυρίως ε, των βιοπραγιών. Και θα ήθελα να σκέφτομαι ότι αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν πρόσφυγες και πέρναγαν τα σύνορα και ερχόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα τους είχαμε ε, καλωσορίσει. Και πολλοί πρόσφυγες που κάνουν το ταξίδι είναι οι άνθρωποι με εξαιρετικές δεξιότητες και γνώσεις και θα πρέπει να τους υποδεχόμαστε στις ε, κοινωνίες μας και στις κοινότητές μας. Για να ενημερώσω τον κύριο Μάθης, κοιτάξτε, την Ευρωπαϊκή Online είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, κάνει ακριβώ αυτό που θέλετε. Και αν υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενδιαφέρον θα το ανακαλύπτατε. Και να καταχωρηθεί ότι ο κύριος Φλίν δεν είναι φεμινιστής καθόλου. Και αν θέλει να γνωρίζει για την ε, φτώχεια όσον αφορά τα ε, είδη υγιεινής των γυναικών να έρθει να μου το πει. Ευχαριστώ Επίτροπε που είσαστε εδώ μαζί μας και όλοι πρέπει να στηρίξουμε, να υποδεχτούμε την πρωτοβουλία που ξεκινήσατε διότι μάλιστα όπως είπατε και τον Ιούλιο θεωρείται ότι είναι τρομοκράτες αυτοί που είναι λαθρέμποροι των πολιτισμικών αγαθών. Και είπατε ότι είναι δουλειά της Ευρώπης να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά. Μου δημιουργούνται δύο ερωτηματικά. Ίσως να δώσετε λεπτομέρειες. Πώς η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ θα παρεμποδίσει τη διασυνοριακή απάτη και σε ποιο δραστήριο επίπεδο χρειάζεται σωστός χρονισμό τη νομοθεσία. Να συντονιστεί με το επόμενο έτος που θα είναι Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Να δούμε ποια είναι η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και από οικονομική πλευρά. Η πολιτιστική κληρονομιά παίζει θεμελιώδη ρόλο. Θετικά να τα δούμε τα πράγματα. Μας διαβεβαιώνεται ότι ο προπολογισμό για προγράμματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά θα είναι προπολογισμό που θα αυξηθεί και δεν θα μειωθεί, όπως είδαμε επί σειρά ετών. Έτσι, να δημιουργούνται ευκαιρίες και για αποκατάσταση και συντήρηση α, της ιστορίας στις χώρες μας. Δεν είναι μόνο να σταματήσουμε το λαθρεμπόριο πολιτιστικών αγαθών και να καθορίσουμε ε, επακριβώς ποια είναι αυτά και να κλείσουμε τα κενά, αλλά και να δραστηριοποιηθούμε, να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στην απόλαυση και συντήρηση της ιστορίας και του πολιτισμού στις χώρες μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Χριστίνα Λιμπάτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε Ήθελα να ξανασυζητήσουμε για το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών ως πηγή χρηματοδότησης του ISIS. Διάβασα μια έκθεση όπου αναφέρεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη πηγή χρηματοδότησης του Ισλαμικού κράτους, τη δεύτερη σημαντικότερη πηγή. Αντιλαμβανόμαστε πόσο ευρύ είναι το πρόβλημα λοιπόν. Όταν υπάρχουν λοιπόν αυτό ως πηγή σημαίνει ότι κάποιος αγοράζει αυτά τα αγαθά. Ποιοι τα αγοράζουν. Πελάτες ε, στο διαδίκτυο για τους οποίους μίλησε ο πρώην Υπουργός Δογεύσκη άνθρωποι που αναζητούν, πώς να το πω, να βρουν έναν τρόπο να, ε, να περάσουν αυτά τα, εργαλεία, τα, τα είδη ε, στις χώρες τους. Ε, σε μια συνεδρίαση με την Ευρωπόλ είχαμε ε, σκεφτεί να πάμε να ελέγξουμε τα ιστοσελίδες αυτές όπου πολλούνται έργα τέχνης, έργα τέχνης τα οποία ενδεχομένως να αγοράζονται με τρόπο παράνομο από κάποιους. Ε, μια ιστοσελίδα όπου να μπορούμε να εντοπίσουμε ενδεχομένως παρανόμως εξεχθέντα ε, ε, πολιτιστικά αγαθά. Καλό θα ήταν λοιπόν να εντοπίσουμε τα αντικείμενα αυτά που αποτελούν το αντικείμενο παράνομου εμπορίου ώστε να μην μπορούν να απολυθούν. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι ο Επίτροπος πρέπει να φύγει σύντομα. Μου είχε πει ότι θα μπορούσε να μείνουν στις 10.30, αλλά από ό,τι φαίνεται πρέπει να φύγει τώρα. Γι' αυτό πολύ σύντομα, Λουίτζι και η Χέλγα Τρίπελ μου είπε ότι δεν έχει απαντήσει στην ερώτησή της. Πολύ σύντομα, Λουίτζι. Ευχαριστώ. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, ευχαριστούμε για την πρόταση. Είναι σαφές κύριε Επίτροπε ότι είναι περιορισμένο το εύρος ε, εδώ της συζήτησης αλλά είπατε τα σημαντικά. Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τομέας αυτός ε, εδώ και έχω να σας ρωτήσω τα εξή. Προβλέπετε κάποια παρακολούθηση αφού μιλάτε πολύ συγκεκριμένα για τα τελωνία. Προβλέπετε κάτι ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν τεράστια κενά στη σχέση μεταξύ αρχών, αρμόδιων υπουργείων κτλ. Ε, θα πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτή την ύπαρξη κενών. Ε, η δεύτερη μου ερώτηση ε, σχετίζεται με το ότι εφόσον θεωρείτε εσείς ότι θεωρείτε ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση, κατάρτιση του προσωπικού ε, που ασχολείται με τα θέματα. Τρίτον, ναι, συμφωνώ να έχουμε γρήγορη έγκριση, αλλά αφού πρόκειται για κανονισμό θα περάσει από το Συμβούλιο, οπότε αναφέρθηκε και η συνάδελφος Σιλβία Κώστα στα ηλεκτρονικά βιβλία. Ναι, θα κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε φυσικά, αλλά μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες τελευταία στιγμή ε, στο Συμβούλιο ε, και τέλος ε, με αυτά που είπατε για τις αρμοδιότητές σας και όλα αυτά ε, οτιδήποτε γίνεται σε αυτόν τον τομέα έχει σημαντικές επιπτώσεις οπότε σας κάνω μια έκκληση ε, για τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιήσετε εσείς Θα είδατε κύριε Επίτροπε πόσο χαιρόμεθα που είστε εδώ και πόσο θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας Σας παρακαλώ λοιπόν σύντομα τον λόγο ε, όσο μπορείτε παρακαλώ απαντήστε σε όλα τα θέματα που τέθηκαν Με τα χαράς να επανέλθω θα με προσοχή τα θέματα. Ο πολιτισμός ε, είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχω πονδύσει πολλά προσωπικά στην δημόσια ζωή μου. Πρέπει να παρουσιάσω, βλέπετε, τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε κάποια λεπτά ε, για κάθε μία από τις χώρες σας. Υπήρξε κάποια παρεξήγηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, πρέπει να κινηθώ προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν και πιο ενδιαφέροντα θέματα βέβαια και πράγματα να κάνουμε. Καταρχάς, θα ήθελα να επιμείνω λέγοντας ότι όλοι καλούνται να συμμετάσχουν στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση που έχει προετοιμαστεί προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έρευνα ήταν διαθέσιμη στο διαδίκτυο επί Λάβαμε απαντήσεις που ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες πολίτες, επιχειρήσεις, ενώσεις, κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές κλπ. Και άλλοι μάλλον και επιλέξαμε προσεκτικά την περίοδο των 250 ετών που είναι αυτό που είχε συμφωνηθεί α, διεθνώς. Γιατί το λέω αυτό. Ποια είναι η ιδέα του κειμένου. Να μην ε, ε, εξετάσουμε αρνητικά τους εμπόρους αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Είναι μια δραστηριότητα που είναι χρήσιμη για τον τομέα, τον καλλιτεχνικό πρέπει να συμμορφώνονται οι νόμιμοι μπορούνε με την ε, εξαγωγή ε, των αγαθών αυτών. Δεν θα υπάρχει μεγάλος αντίκτυπος από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι συμμορφούνται ε, όταν εισάγονται αυτά τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που εστιαζόμεθα είναι εισαγωγή, εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών που γίνεται παράνομα. Και η πρότασή μας έχει προσεκτικά στοχοθετήσει αυτό το τομέα περιμένουμε να αλλάξει η νοοτροπία των αγοραστών που θα μάθουν να περιμένουν από τους εμπόρους των αγαθών κάποια απόδειξη της προέλευσης, ούτως ώστε να φαίνεται ότι είναι νόμιμη η πώληση του αγαθού. Βέβαια, κάποιες ερωτήσεις αφορούσαν πέραν τη, τα, ήταν πέρα των ορίων της προτάσεως για τον προϋπολογισμό και για τους πρόσφυγες εκτός της αρμοδιότητάς μας. Θα επιμείνω επί του ΦΠΑ κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε σειρά προτάσεων. Μείωση ποσοστού ηλεκτρονικά βιβλία. Πρόταση για ΦΠΑ σε δυσονικό επίπεδο. Θέλουμε να έχουμε ένα οριστικό καθεστώς να καλύψουμε τα κενά που επιτρέπουν τις απάτες. 160 δις σε έχουμε και 50 δις για τις απάτες από ΦΠΑ όσον αφορά τις συναλλαγές της διασυνοριακές. Και στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη όσον αφορά το ΦΠΑ. Στο βαθμό που δεν επηρεάζει την εσωτερική αγορά αυτό. Προσεκτικά θα παρακολουθούμε τα τελωνία, σωστά το λέτε, να μην υπάρχουν κενά όσον αφορά το σύστημα, η πρόταση δεν, δεν εξετάζει την επιστροφή παράνομα εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών. Η επιστροφή των αγαθών στη χώρα προέλευσης διενεργείται μέσω διπλωματικών επαφών με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής εκεί που βρίσκονται ε, σε διαπραγματεύσεις μεταξύ της χώρας που βρέθηκαν τα αγαθά και της χώρας προέλευσης. Εργαζόμαστε σκληρά για να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες των τελωνιακών αρχών αυτή η πρόταση επίσης προβλέπει ενίσχυση και καλύτερη κατάρτιση των αξιωματούχων των τελωνίων. Αυτές είναι σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ εκ νέου που μου διαθέσατε τον χρόνο σας. Ήταν προνόμιο για μένα να είμαι παρόν εδώ και βασίζομαι σε εσάς Είδα ότι θα με υποστηρίξετε. Έχετε, δείχνετε υποστήριξη για ταχεία έγκριση της προτάσεως για να εφαρμοστεί γρήγορα και να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών και να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που έχουμε στον τομέα το πολιτιστικό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, χαιρόμαστε και ευχαριστούμε που ήρθατε να βρεθείτε μαζί μας σήμερα εδώ, να μας παρουσιάσετε την πρότασή σας, να απαντήσετε σε ερωτήσεις ε, για τα διάφορα θέματα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσει το νομοθέτημα αυτό από το Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν. Θα... Ελπίζουμε να το μπορέσουμε να το διεκπαιρώσουμε γρήγορα και επιτυχώς. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα.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 Λοιπόν, είναι εδώ όλοι οι εμπειρογνώμονέ μα. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη. Αυτή τη συνεδρίαση εργασία για την πολιτιστική δουλειά με τους πρόσφυγες που οργάνωσε το τμήμα πολιτικής μας. Έχουμε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες που ήρθαν στην Ευρώπη το 2015. Οπότε οι κοινωνίες υποδοχής ε, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις για να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η συνεδρίασή μας θα δει και θα εξετάσει πώς μπορεί να βοηθήσει η πολιτιστική δουλειά με τους πρόσφυγες στην υπέρβαση αυτών των προκλήσεων και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει. Έχουμε μια σειρά από εμπειρογνώμονες που θα μας βοηθήσουν ε, ε, να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε την καθηγήτρια Alison Phipps του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Έχει την έδρα UNESCO για την ένταξη των προσφύγων μέσω της ε, εκμάθησης γλωσσών και των τεχνών. Είναι συντονίστρια του δικτύου της Γλασκόβης για το άσυλο και την μετανάστευση. Θα μας μιλήσει για αυτά τα θέματα. Έχουμε την κυρία Νεζούγα Φρόσερ που είναι στην ε, ε, υπεύθυνη για τους ίδιους ε, τομείς και εργάζεται στην ε, ε, Γλασκόβη μαζί με την κυρία Φίπς και θα μας δείξει πολύ συγκεκριμένα, όπως θα καταλάβετε όλοι, τι αποφασιστικό ρόλο παίζει η συνεργασία και οι διαπολιτιστικές επαφές στην προσπάθεια αυτή. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε με μεγάλη αναμονή ε, αυτά που θα μας πούν έχουμε και τον Ρασούλ Νεάντμε που είναι υπεύθυνο για τα πολιτιστικά θέματα στην περιοχή Βέστρα Γκέτελαντ και εκπροσωπεί την Σουηδία στην ομάδα εργασίας των κρατών μελών για, την, για τον διαπολιτισμικό διάλογο. Θα ασχοληθεί με θέματα της σημερινής πρακτικής της δουλειάς με τους πρόσφυγες και τι διδάγματα μπορούμε να εξάγουμε. Επίσης καλωσορίζω την Ροζάνα Λούις έχει ασχοληθεί με θέματα της προώθησης του πολιτισμού είναι πολυμαθής, έχει πολύ συγκεκριμένη εμπειρία από το καταβλισμό προσφύγων στο Καλέ και έναν άλλο καταβλισμό στην Κοπενχάγη και έχει ασχοληθεί με την υποστήριξη των προσφύγων μέσω της επόμενης γενιάς των προγραμμάτων της Ένωσης. Κάθε εμπειρογνώμονας μας έχει 10 λεπτά και τους παρακαλώ να μην υπερβούν τον χρόνο τους γιατί θέλουμε να συζητήσουμε. Να μας μείνει χρόνος για ερωτήσεις. Καταρχάς, να δώσω το λόγο στην κυρία Φίπς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση να συμβάλλω σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Με λένε Άλισον Φίπς και είμαι στην πρώτη θέση, στην, για πρώτη φορά προεδρία όσον αφορά τις πρόσφυγες ε, και την ένταξη των προσφύγων μέσω των γλωσσών και των τεχνών. Αυτή είναι η δομή της παρουσιάσεως μου. Θα παρουσιάσω το προβληματισμό που παρουσιάζεται από τις διάφορε μελέτε τις πανεπιστημιακές. Θα δώσω παραδείγματα για το πώς, πώς οι διάφορες ιστορικές, τα ιστορικά σχήματα για την εκπροσώπηση και παρουσίαση των προσφύγων επαναλαμβάνονται και εμποδίζουν την πολιτιστική τους ένταξη στην κοινωνία και την ευημερία τους. Θα παραθέσω παραδείγματα πολιτιστικών εργασιών υπό έναν τίτλο που περιγράφει διάφορα είδη εργασία στον πολιτιστικό τομέα, δίνοντας παραδείγματα που γνωρίζω από όλο τον κόσμο και που σε κάποιες περιπτώσεις έχω εμπειρία άμεση και πρακτική εμπειρία και μετά θα προβώ σε συγκεκριμένες ε, συστάσεις. Λοιπόν, πώς μπορούμε να δούμε το πολιτιστικό έργο με τους πρόσφυγες μέσω καλλιτεχνικών προγραμμάτων, κοινοτικών προγραμμάτων που παρουσιάζουν τη ιστορία των προσφύγων ή παρουσιάζουν εικόνες και επιδόσεις ε, και παραστάσει των προσφύγων και σε κάποια περίπτωση ε, με τη συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων. όμω. η πιο επιτυχη χρήση καλλιτεχνικών ε, ε, αισθητική παρουσίαση των έργων των προσφύγων είναι για λόγου προπαγάνδας που δεν διευκολύνουν την ένταξη αλλά την απομόνωση και δεν προωθούν την ένταξη και πολύ συχνά προωθούν συγκεκριμένο θεματολόγιο για θέματα ασφαλείας. Υπάρχουν δύο σημεία που πρέπει να παρατηρήσουμε αυτή τη διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα, τη χρήση μιας γλώσσας που βγάζει τον ανθρώπινο παράγοντα από την περιγραφή. Περιγράφει τους πρόσφυγες με έναν τρόπο σαν ορδέ, σαν, με έναν τρόπο που δεν έχει τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Και είναι στο βαθμό 6 6 ε, στους 10 βαθμούς του Ινστιτούτου Γενοκτονίας είναι η περιγραφή. Δηλαδή που υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να γλιστρήσουμε προς μια συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενοκτονία. Ε, είναι πολύ σοβαρό θέμα, δηλαδή τρόπος παρουσιάζονται. Μετά, η ανακύκλωση εικόνας και αφηγημάτων της ιστορίας που μπορεί να έχει ξεκινήσει πολύ παλιά. Βλέπετε στη διαφάνεια εικόνες που ξεκινάνε από την εκστρατεία του Brexit και φτάνουν στο ολοκαύτωμα ε, που ιστορικά ε, αναφέρονται και οι πρόσφυγες οι Ουγγενώτοι Και όλα αυτά οδήγησαν σε μια αύξηση του φόβου για τον ξένο και κυρίως για τους πρόσφυγες όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία. Ε, πολιτιστική δουλειά αυτού του είδους έχει τροφοδοτήσει αυτή την, αυτό το φόβο διονύζοντας αυτές τις εικόνες και αυτή την διατύπωση και την γλώσσα που επαναλαμβάνεται στην ιστορία. Η δεύτερη πιο ε, κοινή χρήση πολιτισμικού έργου με τους πρόσφυγες είναι να χρησιμοποιούν τους ε, στόχους ένταξης και υποδοχής. Δηλαδή να δείξουμε πώς υποφέρουν οι πρόσφυγες. Ε, ηγούνται κυρίως οι καλλιτέχνες αυτή την προσπάθεια, ε, δείχνουν κάποιες κατευθύνσεις και θέλουν να αλλάξει η νοοτροπία, να υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή από όλα τα, από όλα τα μέρη της κοινότητας. Επίσης χρησιμοποιείται από ΜΚΟ σαν ένα όχημα για τη συλλογή χρημάτων και υποστήριξη των αποστολών των ΜΚΟ. Λοιπόν, πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτά τα σχήματα, τα στερεότυπα της ιστορίας. Εδώ σας παραπέμπω στην προσπάθεια τη ρηξικέλευτη από την Αυστραλία, του RISE. Είναι μια, ένα, ένας οργανισμός τον οποίο ηγούνται οι πρόσφυγες και το μανιφέστο τους για προθή έργα τέχνης και πολιτιστικό έργο. Κάτι που υιοθέτησα και εγώ για τους πανεπιστημιακούς. Το RISE τονίζει τα εξή. Το πολιτισμικό έργο με τους πρόσφυγες δεν είναι κάτι ουδέτερο. Οι πρόσφυγες είναι φορείς δεν είναι παθητικοί ευγνώμονες αποδέκτες. Οι πρόσφυγες πρέπει να προσεγγιστούν με κρίσιμο όμα, μια στάση ε, αυτογνωσίας αν θέλετε. Και η τέχνη που παράγεται για την τέχνη και ότι αυτό που είναι καλό για τους πρόσφυγες δεν είναι απλώς κάτι λειτουργικό, θα είναι κάτι καλό για όλους. Λοιπόν. Δεν είναι εύκολο σαν Αφρικανός μετανάστης να διακόψει έναν καθηγητή της μεσαίας τάξης, λευκό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα έργου του πολιτιστικού τομέα με συνεργασία για τους πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες που θα πρέπει να εξεταστούν και ληφθούν υπόψη. Το πρώτο είναι ένα παράδειγμα ενός θεάτρου που χρησιμοποιήθηκε από την ύπατη αρμοστία του Ι.Ε. για τη μέρα των προσφύγων φέτος. Τι πήραν μαζί τους ήταν ο τίτλος και διασημότητες συμμετείχαν, χρησιμοποιούν ε, τη γλώσσα για να μας συγκλονίσουν από, ε, από την υπνηλία μας. Πήραμε την παρθένιά μας στη θάλασσα, παράδειγμα. Ε, ανοιχτήκαμε με μετότος ώστε οι πειρατές να μην μας αγγίξουν. Αυτό ευαισθητοποιεί τον κόσμο και δείχνει τις συγκλονιστικές εμπειρίες κυρίως γυναικών και κοριτσιών ε, χωρίς να υπάρχουν ε, ανθρωπιστικοί διάδρομοι και δείχνει ποιες είναι οι συνέπειες του κλεισίματος των συνόρων. Αυτά είναι τα διαμερίσματα Red Road Flats στη Γλασκόβη. Αυτό το έργο πήρε στέγαση που χρησιμοποιείται για τον τόπιο πληθυσμό και για τους ετούντος άσυλο μαζί, αλλά είχε προβλήματα υγείας και υγρασίας και μετατρέπει σε ένα χώρο για ανάμνηση, για θρήνο και ανασυγκρότηση πριν καταστραφεί. Ε, συνελέγησαν τραγούδια που τραγουδούσαν τα παιδιά ε, στα διαμερίσματα και τα παίξαν από μεγάφωνα σε πολλές γλώσσες. Και τελικά έγιναν τελικά ένα τεράστιο μεγάφωνο για να το ακούει όλη η πόλη αυτό το κτίριο. Ε, τα, παιδιά ε, έδειξαν και παρουσίασαν χρώματα που τα συνέδεαν με τις πατρίδες τους και χρωμάτισαν σεντόνια τα οποία τα κρέμασαν από τα παράθυρά τους και ε, μάζεψαν επίσης και θηβετιανές σημαίες προσευχής και ετοίμασαν έτσι εκ του προχείρου μια χοροδία που τραγούδισε ένα αποχαιρετιστήριο. Και τώρα είδαμε εδώ το νέο ε, βιβλίο με διάφορα τραγούδια και στίχους, συνεργασία του Διεθνούς Φεστιβάλ του Εδιμβούργου και του Βρετανικού Συμβουλίου με το BBC Arts. Μαζέψαμε διάφορες καλλιτέχνες από την Global South, την Άντεν Σουα Τότζο που είναι εδώ μαζί μας, και βοηθούν όλοι αυτοί την ένταξη των προσφύγων μαζί με την Καρίν Πολ που είναι βασική τραγουδίστρια folk της Κορτίας και ετοίμασαν νέα δουλειά μαζί συγχωνεύοντας παραδόσεις, ρυθμούς, αρμονίες με ένα μουσικό βίντεο το οποίο τον εμπνεύστηκαν από αυτά που έπαθε ο Ελάν Κούρντι, πρόσφυγος, που ξεβράστηκε στις παραλίες της Τουρκίας. Θέλουμε να σπάσουμε ε, τα διάφορα στερεότυπα της ιστορίας που ήταν τοξικά για τη μνήμη μας. Ένας λευκός επαγγελματίας με ε, κουστούμι είναι αυτός που ζητά βοήθεια. Χρειάζεται βοήθεια. Είμαστε όλοι πρόσφυγες, όπως είπε η Χάνα Αρέντ. Κάπου είμαστε πρόσφυγες όλοι. So Και τελικά πάω στις συστάσεις μου. Ε, πενώ ε, αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Θα έπρεπε οι κατευθύνσεις γραμμές του ΡΑΙΣ σε μελλοντικά μέτρα να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να εστιαστούμε επί προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνουν τους πρόσφυγες που αφορούν την ένταξη και πολυγλωσσική δραστηριότητα. Επενώ την χρήση πολλών ε, πράξεων δημιουργικότητας τοπικών κοινοτήτων που βασίζονται σε νέες σχέσεις που προωθούν τη φροντίδα για καινοφανείς δραστηριότητε και πράξεις μαρτυρίας, καταγραφής και υπόμνησης κοινωνικών αλλαγών. Τέλος, θα ήθελα να επεκταθώ λίγο στην έρευνα και τη μαρτυρία που αποδεικνύουν ότι το πολιτιστικό έργο για διαπολιτισμική ευημερία με τους ε, πρόσφυγες είναι κάτι που είναι πιο αποτελεσματικό για το κοινό ε, αγαθό, για, για το κοινό καλό όλων, όταν θυμάται, ε, θρηνεί, βοηθά την αμοιβαία αποκατάσταση, παρουσιάζει την αλήθεια για την ανθρώπινη κατάσταση και επίσης είναι μια δραστηριότητα στην οποία είναι χαρά να συμμετέχει κανείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φίλιπς Κυρία Φίλιπς, μάλλον, συγγνώμη. Και ευχαριστούμε θερμά. Την... Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που είχαμε τέτοια παρουσίαση εδώ και ήταν πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό και συμπαθητικό. Και τώρα έχουμε τον κύριο Μερ και τον παρακαλώ ε, να κάνει την παρουσίασή του 10 λεπτά και εκείνος. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Ε, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ για να σας ε, μιλήσω εκ μέρους ε, των ε, μεταναστών σαν εμένα να σας πω ότι ένα από τα δώρα που προσφέρει η σημερινή προσφυγική κρίση είναι ότι οδήγησε σε πάρα πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες και πολιτισμικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να ταξινομήσει κανείς εύκολα τόσες πολλές δραστηριότητες. Θα προσπαθήσω ωστόσο να ε, προσδιορίσω κάποια μοτίβα, κάποιες δομές ε, που θα τις κάνουν πιο κατανοητές τους ανθρώπους οι οποίοι έμεσα ή άμεσα ε, μπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην δομή της παρουσίασής μου που είναι και η δομή του εγγράφου μου ε, εξετάζουμε καταρχάς τους διάφορους τύπους ε, προγραμμάτων, τις διάφορες ε, προσεγγίσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Στη συνέχεια θα δούμε την κοινωνία των πολιτών, πώς δείχνουν τεράστια αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και μετά το κοινό καλό που προκύπτει από την πολιτιστική συνεργασία των κοινωνίων των πολιτών με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και τέλος θα εστιαστώ στα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από τη συνεργασία με τους πρόσφυγες. Όταν μιλάμε τώρα για διάφορους τύπους ε, προγραμμάτων, εκεί ρωτάμε το βασικό ερώτημα ποια είναι η σχέση ε, ε, εξουσίας ουσιαστικά εντός του κάθε προγράμματος, ποιος κυριαρχεί, ποιος ηγείται και, ποιος, και ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για την επιτευξή των στόχων. Βασί των ερωτημάτων αυτών έχω εντοπίσει πέντε τύπους έργων. Τα ήδη έτοιμα, τα οποία παραδοσιακά, τα κλασικά ε, προγράμματα που έχουν ήδη σχεδιαστεί για τους ε, πρόσφυγες χωρίς αυτοί να έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό. Τα έργα που έχουν σχεδιαστεί από κοινού με τους πρόσφυγες, τα co-design, το, στη ε, δεύτερη κατηγορία, τα συμμετοχικά επίσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί μόνο από πρόσφυγες ε, ώστε να ενδυναμωθούν στο πλαίσιο κάποιες οργάνωσης, τα διατομεακά επίσης, τα οποία δεν κάνουν διαχωρισμό εθνότητας, μάλλον κάνουν τέτοιο διαχωρισμό, αλλά μόνο ως ενός χαρακτηριστικού μεταξύ πολλών άλλων. Και μετά έχουμε ε, τα διατομεακά στην πέμπτη κατηγορία, που περιλαμβάνουν πολλούς τομείς ε, σε μια κοινωνία. Τώρα, όταν μιλάμε για τα κράτη-μέλη, εδώ εστιαζόμαι σε δύο κατηγορίες ε, κρατών μελών. Τα κράτη πρώτης γραμμής, όπου, από όπου εισέρχονται οι πρόσφυγες, ε, εκεί η εστίαση, το βασικότερο ζήτημα είναι να, παρέχεται, να παρέχονται στους πρόσφυγες ε, τα βασικά κάποιες δραστηριότητες που να τους απασχολήσουν μέχρι να κινηθούν ε, στην κέντρο της Ευρώπης. Μετά έχουμε τις χώρες υποδοχής όπου υποβάλλουν ε, αίτηση ε, μόνιμης διαμονής οι πρόσφυγες. Εκεί το θέμα είναι η πλήρης ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία και εκεί έχουμε δύο προσεγγίσεις. πρώτη βλέπει την, την πολυπολιτισμικότητα ως μια ενδιάμεση κατάσταση, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να λήξει το συντομότερο δυνατόν. Και εδώ τα έργα ουσιαστικά είναι φιλανθρωπικά. Η άλλη προσέγγιση αφορά τις χώρες που θεωρούν την πολυπολιτισμικότητα και την μετανάστευση ως κάτι φυσιολογικό. Μια φυσιολογική πτυχή της σημερινής, της σύγχρονης ζωής και της κοινωνίας. Εδώ λοιπόν αυτές οι κοινωνίες εστιάζονται περισσότερο στην ε, χειραφέτηση, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη συμμετοχή. Ε, ψάχνουν να δουν πώς μπορεί ο πρόσφυγας να γίνει ε, πλήρες μέλος της ε, κοινωνίας. Τώρα, όσον αφορά εδώ τι δράσει τη κοινωνία των πολιτών, εστιάζομαι σε δύο πτυχέ. Πρώτον, στην οικουμενική φιλοξενία βασισμένο στα λόγια του Εμμανουέλ Καντ, ενό από του προπάτορε του ευρωπαϊκού μοντέλου. Η ιδέα εδώ είναι ότι έχουμε έναν ενιαίο πλανήτη, τον οποίο πρέπει να προστατεύουμε σε δύσκολε στιγμές. Με άλλα λόγια, χρωστάμε φροντίδα ο ένας τον άλλο. Η άλλη πτυχή στην οποία εστιάζομαι είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να δραστηριοποιούνται περισσότερο ε, σε θέματα οργάνωσης της κοινωνίας ε, για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Και μια πτυχή αυτού είναι ε, οι δημόσιες αξίες που χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αξιολόγησης ε, των αποτελεσμάτων ε, των κοινωνιών αυτών όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων. Στην επόμενη διαφάνεια ε, μιλάω για τα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από τη σημερινή προσφυγική κρίση. Η πρώτη έχει να κάνει, το πρώτο έχει να κάνει με τη χειραφέτηση των προσφύγων, επειδή είναι ένα ζήτημα που όλο ένα συζητάμε στα διάφορα έργα. Εδώ βασίστηκα στην ιδέα ότι η χειραφέτηση σημαίνει πολιτική συμμετοχή μαζί με όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Να μπορεί δηλαδή να συμμετέχει κανείς με το δικό του τρόπο ζωής ε, στα κοινά. Το άλλο δίδαγμα αφορά την κοινωνική κινητικότητα. Εδώ η έρευνά μου και η ανάλυση μου βασίστηκαν στο γεγονός ότι πολλά έργα αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τον όρο ένταξη, το integration, διότι φαίνεται να στιγματίζει αντί να βοηθά τους ε, πρόσφυγες. Η κοινωνική κινητικότητα είναι μια γενικότερη έννοια που καλύπτει όλες τις δυνατότητες ε, βελτίωσης της ζωής ε, των προσφύγων σε κάθε κοινωνία, αντί να μένουν κολλημένοι στη θέση του πρόσφυγα, του αδύναμου πρόσφυγα. Το επόμενο δίδαγμα αφορά το πώς μπορούμε να ε, συνδέσουμε ε, τα ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες ε, με τα ζητήματα που αφορούν τον πληθυσμό φιλοξενία, ώστε να μην δημιουργούνται εντάσει. Ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πρόσφυγε δεν βρίσκονται εδώ για να καταστρέψουν τα κοινωνικά συστήματα, αλλά να συμβάλλουν τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Σε αυτή τη διαφάνεια τώρα εδώ βλέπετε τα συμπεράσματά μου. Τα πολιτισμικά έργα χαρακτηρίζονται και από επιτυχίε και από αποτυχίε. Επιτυγχάνουν όταν βασίζονται σε ανθρώπινα δικαιώματα, είναι συμμετοχικά, είναι διαπολιτισμικά, διατομέακα ε, και οριζόντια και αφορούν ζητήματα που απασχολούν και τους πρόσφυγες και τους πληθυσμού φιλοξενία. Αποτυγχάνουν όταν παρασμένουν εντό ορισμένων κλασικών κλειστών ορίων ε, εθνικών ταυτοτήτων και πολιτισμών. Τέλος, έχω κάποιες συστάσεις, δύο σύνολα συστάσεων, ε, ένα σύνολο για τους ε, ενδιαφερομένους και ένα για όσους χαράσουν πολιτική. Πρέπει να ενθαρρύνονται τέτοια έργα, ε, έργα τα οποία βασίζονται σε ανθρώπινα δικαιώματα, που χειραφετούν τους πρόσφυγες σε δομικό επίπεδο, που έχουν ίση συμμετοχή προσφύγων και τοπικών πληθυσμών, και που καταπολεμούν το ρατσισμό, το σεξισμό, τον εξτρεμισμό και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και τα οποία είναι οριζόντια και διατομεακά. Αφορούν δηλαδή όλους τους τομείς. Συνιστώ ιδιαίτερως ε, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και ειδικότερα των οργανώσεων που δημιουργούν οι ίδιοι οι πρόσφυγες ώστε, για, για παράδειγμα τις ε, διαδικασίες ε, αίτησης χρηματοδότησης. Η επόμενη σύστασή μου είναι να ενσωματωθούν κριτήρια συμμετοχής και μηχανισμοί αξιολόγησης ε, στα κριτήρια χρηματοδότησης. Και τέλος, για να υπάρξει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και εθνικών και διεθνικών επιπέδων, καλό είναι να συνδεθούν τα έργα αυτά ε, που αφορούν τους πρόσφυγες ε, με ένα γενικότερο αφήγημα ε, περί κάποιου κοινού οράματος για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τη δική σας παρουσίαση. Οι κυρίες Λούις και Μάρτιν, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Δέκα λεπτά και εσείς παρακαλώ για την παρουσίαση σας. Ε, θα το κατανέμετε το χρόνο αυτό μεταξύ σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χαιρόμεθα για τη δυνατότητα που έχουμε να παρουσιάσουμε την ερευνά μας και τα κυριότερα πορίσματά μας για την πολιτιστική εργασία ε, εργασία με τους πρόσφυγες. Ασχολούμεθα με τρία βασικά θέματα. Τι μπορούμε να μάθουμε από τα προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί τώρα, τι γενικές ε, συστάσεις μπορούμε να κάνουμε για τα επόμενα προγράμματα σε αυτό το τομέα και πώς ε, τα συγκεκριμένα πολιτιστικά προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των προσφύγων. Για το πρώτο θέμα, τα πιο σημαντικά και σχετικά προγράμματα είναι το Erasmus η Δημιουργική Ευρώπη και η Ευρώπη για τους πολίτες που είναι εντό ε, των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σας. Και τα τρία έχουν πλευρές που εστιάζουν στην εργασία με τους πρόσφυγες και έχουν πρόσβαση διάφοροι πολιτιστικοί οργανισμοί και πρωτοβουλίες σε αυτά. Το έρασμο ΣΥΝ ε, έχει το θετικό ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις παντού στην Ευρώπη. Και βεβαίως ε, μπορεί να συνεργαστεί με πολιτιστικούς οργανισμούς και για δραστηριότητες που αφορούν τους πρόσφυγες Κανένα από αυτά τα δύο στοιχεία δεν είναι το βασικό ε, στοιχείο του προγράμματος. Οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις του πολιτικού τομέα δεν γνωρίζουν ε, πολύ καλά το πρόγραμμα αυτό. Και οι κυριότερες οργανώσεις που ασχολούνται έχουν ε, ήδη εκαθιδρυμένα ευρωπαϊκά δίκτυα λόγω του διεθνικού χαρακτήρα του προγράμματος. Η Δημιουργική Ευρώπη ε, έχει παίξει πολύ θετικό ρόλο στην εργασία με τους πρόσφυγες. Το 2016 έγινε μια συγκεκριμένη προκήρυξη για τη στήριξη της ένταξης των προσφύγων και έτσι θαρρήθηκαν πολιτιστικές οργανώσεις για να εργαστούν για θέματα προσφύγων. Αλλά κυρίως ασχολείται με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ παρομοίων οργανώσεων στην Ευρώπη. Ε, στηρίζει άμεσα τους πρόσφυγες και, τους, και τις οργανώσεις που τους βοηθούν. Η Ευρώπη για τους πολίτες μπορεί να βοηθήσει μέσω των ε, προγράμματων για την κοινωνία των πολιτών και για τη δικτύωση των πόλεων. Και έτσι ε, βοηθάει προγράμματα που είναι πιο βαθιά ριζωμένα και η ηγεσία τους είναι από τις τοπικές κοινωνίες και συνδέει την κοινωνία των πολιτών και τις ε, ενωσιακές πολιτικές για να υπάρξει διάλογος και για να υπάρξει περισσότερη ορατότητα των προγραμμάτων της. Αλλά ε, δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την ευρύτητα των θεμάτων και τον αριθμό των οργανώσεων που θέλει να στηρίξει. Αυτό περιορίζει τον αριθμό των προγραμμάτων για την πολιτιστική δουλειά με πρόσφυγες που μπορεί να βοηθήσει. Και τώρα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο την ε, Πόλη που θα μας μιλήσει για την ε, εμπειρία μας με τα προγράμματα αυτά. Είχαμε συζητήσεις με τα διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και γενικά εκτιμά τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα τη δυνατότητα συνεργασίας με παρόμοιες οργανώσεις ε, από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αλλά υπήρξαν διάφορες ανησυχίες για τα εξή σημεία. Πρώτον, κατά πόσο βοηθάμε να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι ίδιοι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες πολλές φορές αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα, ενώ έχουν πολύ διαφορετική προέλευση, γλωσσική, πολιτιστική, και γι' αυτό είναι σημαντικό τα προγράμματα να βοηθούν του πρόσφυγε να αναλάβουν ίδιοι πρωτοβουλίε. Να λάβουν υπόψη λοιπόν και τι ατομικέ και τι συλλογικέ ανάγκε των προσφύγων πριν του ε, φέρουν σε επαφή με τι τοπικέ κοινωνίε. Η καλύτερη συμπερίληψη από την αρχή των προσφύγων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων παίζει καλό ρόλο. Η ένταξη είναι, δεν είναι μονόδρομος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να βοηθήσουμε περισσότερους ασφαλείς χώρους για να γίνεται διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες των προσφύγων, και να υπάρξει ε, ενίσχυση της αλληλοκατανόησης και καλύτερη κατανόηση των αναγκών των προσφύγων. Επίσης, τα αποτελέσματα πρέπει να γίνονται ευρύτερα γνωστά. Αυτό θα βοηθήσει τα μελλοντικά προγράμματα, τα επόμενα προγράμματα. Θα καταλάβουμε ποια ήταν τα θετικά και αρνητικά των ε, προηγούμενων προγραμμάτων. Θα γίνεται καλύτερα αξιολόγηση. Θα υπάρχει πιο διαφανή συνεργασία. Οι μικρότερες και τοπικές οργανώσεις ε, πολλές φορές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες που έχουν ε, καλύτερες δυνατότητες για να αναλάβουν το διοικητικό άχθος ενός προγράμματος και μπορεί να λαμβάνουν και από αλλού χρηματοδότηση. Χρειάζεται περισσότερη προχρηματοδότηση και συμπερίληψη μικρότερων οργανώσεων στα προγράμματα. Αυτό θα οδηγούσε σε καλύτερες συνεργασίες. Επίσης προτάθηκε ότι η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να δίδεται μόνο σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε χώρες που έχουν εταιρική σχέση, αλλά και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα χώρες της Μέσης Ανατολής και της νότια Αφρική. Αυτό θα άνοιγε πολιτιστικά σύνορα και θα οδηγούσε σε μια πολυτομιακή προσέγγιση. Και τώρα η Ροζάνα θα σα παρουσιάσει τις κύριες συστάσεις μα. Λοιπόν, όπω ήδη είπαμε, χρειάζεται να αυξηθεί το επίπεδο χρηματοδότηση και για τα τρία προγράμματα, ιδιαίτερα για πρωτοβουλίε που αφορούν την πολιτιστική δουλειά για του πρόσφυγες. Χρειάζεται περισσότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να αγγίξουμε ένα ευρύτερο ακροατήριο, ούτω ώστε περισσότερα άτομα από πολύ διαφορετικές προελεύσεις ε, να ωφεληθούν. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη δικτύωση, ε, είτε ε, φυσική είτε μέσω του διαδικτύου, θα βοηθήσουν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να απλοποιήσουμε την διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Είναι πολύ περίπλοκες και βαριέ για πολλέ οργανώσει αυτέ οι διαδικασίε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα όπου όσοι, έχουν, όπου όσοι ήδη έχουν λάβει χρηματοδότηση και έχουν ολοκληρώσει προγράμματα να περάσουν την πείρα του και την ε, ομότιμη εκπαίδευση, την εκπαίδευση μεταξύ ομοτήμων δηλαδή. Αυτές οι ανταλλαγέ θα βοηθούσαν πολλού να υποφεληθούν από τη χρηματοδότηση και θα αύξαναν και την ποιότητα των προγραμμάτων. Η πολιτιστική δουλειά με τους πρόσφυγες έχει διαφορετικές μορφές. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις λεπτομέρειες, να δούμε τι ακριβώς επιδιώκουμε, τι αποτελέσματα θέλουμε. Αυτά πρέπει να τα ορίσουμε καλύτερα για να καταδειχθεί ε, κατά πόσο και με τι τρόπο ωφελούνται και οι πρόσφυγες και οι κοινωνίες υποδοχής. Στην επόμενη φάση προγραμματισμού πρέπει να συλλέξουμε πολύ περισσότερα στοιχεία για το τι επίπτωση έχουν αυτά τα προγράμματα και ως αποτέλεσμα και ως διαδικασία. Αυτά τα αποτελέσματα πρέπει κατόπιν να γίνουν ευρύτερα γνωστά για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση για το ρόλο του πολιτισμού στην ένταξη των προσφύγων. Επίσης, ε, πρέπει να αναπτύξουμε ένα ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης που να προσαρμόζεται στις ε, φυσικές και κοινωνικές ανάγκες και των προσφύγων και των τοπικών κοινωνιών. Άρα κυρίως θέλουμε να έχουμε ε, προγράμματα προσαρμοσμένα, επιμέτρο, ε, παντού στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν όμιλο προγραμμάτων που να ενδιαφέρονται για την πολιτιστική δουλειά για τους πρόσφυγες, που θα συνεργάζονταν σε όλους τους τομείς για να συμμερίζονται τις βέλτιστες πρακτικές, να βοηθούν την συνειδητοποίηση για να επηρεάσουν την πολιτική και να ε, χρηματοδοτήσουν και προγράμματα που θα ε, ε, προωθούν τη δουλειά από, για και με τους πρόσφυγες. Έτσι θα αναπτύξουμε πολιτιστικά προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες. Το πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε βεβαίω να χρηματοδοτηθεί επαρκώς για μια σημαντική χρονική περίοδο για να έχει μια ε, μακροχρόνια επίπτωση και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και σε ευρωπαϊκό. Η εκθεσή μας δεν εξέτασε τις χώρες της νότιας γειτονίας, αλλά μπορούμε να πάθουμε, να μάθουμε συγγνώμη, πολλά από τη δουλειά με τους πρόσφυγες σε αυτή την περιοχή. Για παράδειγμα, χρηματοδοτήθηκε μία μελέτη για το πρόγραμμα MedCulture, που είναι μία πολιτιστική προσπάθεια πολιετής που γίνεται με τρόπο χωρίς αποκλεισμού και με συμμετοχή των ίδιων των αφορομένων. Βεβαίως, ε, το πρόγραμμα ίσως να μην ε, προσαρμόζεται στις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, αλλά οι δραστηριότητες του βοηθούν πολλούς μέσω συναντήσεων, ε, καταρτήσεων και δύο προγράμματα χρηματοδότησης υποπρογραμμάτων. Προωθεί επίσης την ελευθερία της έκφρασης και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά μας αφορούν ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα για τη δουλειά με τους πρόσφυγες. Καταλήγοντας, ελπίζουμε αυτή η ενημέρωση να σας βοηθάει για τα επόμενα προγράμματά σας τα διδάγματα ε, από τα ολοκληρωμένα και υποεξέλιξη προγράμματα καθορίζουν τα βασικά στοιχεία της δουλειάς με τους πρόσφυγες, εξετάζουν καινοτόμα σχήματα για μετά το 2020. Όπως είπαμε και στην έκθεση για φωνές του πολιτισμού, τα πολιτιστικά προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τη συλλογική πρωτοβουλία των ε, προσφύγων και να τους επιτρέψουν να αποκτήσουν πολιτικό και κοινωνικό βάρος. Ε, Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιτύχουν αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς τις δύο για τις παρουσιάσεις σας και των προτάσεών σας που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Να περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις 50. Να δώσω τον λόγο πρώτα στους συντονιστές, εφόσον θέλουν, και κατόπιν και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Νομίζω ότι θα προλάβουμε. Η Ζαμπίνε Φεχάιν. Ε, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση των μελετών αυτών. Τα πολιτιστικά προγράμματα είναι πολύ σημαντικά για την ένταξη των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Μία ερώτηση. Τι βαθμό αποδοχής έχουν τέτοιες ε, πρωτοβουλίες στα διάφορα κράτη-μέλη. Πόσα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται και προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα κύρια σημεία με τα οποία ασχολείστε. Μπορείτε να μας πείτε ε, πώς ε, κατανέμονται εδαφικά λοιπόν ε, τα προγράμματα αυτά και τι βαθμό αποδοχής, πώς γίνονται δεκτά, πόσες χώρες και σε τι βαθμό πραγματικά ενδιαφέρονται και προωθούν τα κράτη-μέλη την ένταξη μέσω του πολιτισμού. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτές τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Ε, σας συγχαίρω για την επιλογή ε, των ομιλητών ε, και να συγχαρώ και την ε, καλλιτέχνηδα που τραγούδησε. Πιστεύω ότι περνάμε σε μια διαφορετική φάση. Έχουμε ένα δομικό θέμα προκύπτει σήμερα. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη για να μπούμε σε μια δεύτερη φάση ορίμανσης των πολιτικών που γίνονται πιο ευσυνείδητες και με τη βοήθεια διαφόρων ενώσεων προσφύγων που όπως δείξατε εσεί και στη δική μου τη χώρα την Ιταλία αποτελούν πλέον ε, αναπόσπαστο κομμάτι και τη απάντηση. Δεν είναι ότι ένας κάνει προτάσεις ε, μόνο και ε, τρία είναι τα βασικά σημεία. Πρέπει να αλλάξουμε την οπτική γωνία όπως είπατε και εσείς να περάσουμε από μια φιλανθρωπική προσέγγιση σε μια προσέγγιση που να βασίζεται στην αξιοπρέπεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπατε και εσείς κύριε Νετζαντμέρα και πάντα είναι επίκαιρο το θέμα της ε, χειραφέτησης. Αυτό αφορά και τον τρόπο με τον οποίο αφηγούνται την κατάσταση τα μέσα. Βγαίνει λίγο από το θέμα των τεχνών, αλλά εντάστε στον πολιτισμό παρόλα αυτά. Το βλέπω και στη χώρα μου και σε όλη την Ευρώπη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, είναι ο χειρότερος εχθρός των πολιτικών ε, ένταξη. Όπως είπατε, μιλούν για ορδές, ε, για ροές, για κίνδυνο. Και ο μεσός πολίτης στην Ιταλία, για παράδειγμα, αν πάει και δει ποιον ξέρει που επηρεάζει θετικά τη ζωή του, εκεί αλλάζει η οπτική γωνία. Ε, το θέμα αυτό δεν το εξετάζουμε επαρκώ. Πιστεύω ότι μια ισχυρή συμμαχία με τι δημόσιε αρχέ και με, τις τηλεοπτικές, ε, με τους τηλεοπτικούς οργανισμούς και τα μέσα μαζική ενημέρωση είναι θεμελιώδους σημασίας. Δεν έχει νόημα να καθόμαστε, να διηγούμαστε ιστορίες, ε, να... Οι πρόσφυγες μας ξαναδίνουν μια ταυτότητα που ίσως δεν έχουμε χάσει ως αξίες αναφοράς. Κάτι άλλο, υπογραμμίσατε πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματά μας, ε, γιατί και γι' αυτό, με αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε σε αυτές τις κρίσιμες εποχές. Ε, μιλήστε για περαιτέρω προτάσεις, τις έχω δει, αλλά λέτε πρέπει να έχουμε πιο προσαρμοσμένα, πιο ειδικευμένα προγράμματα για το θέμα αυτό. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε πιο λεπτομερώς, διότι εμείς ε, έχουμε προσπαθήσει να εντάξουμε ε, στο Creative Europe και σε άλλα προγράμματα το θέμα αυτό, ίσως ανεπαρκώς πώ θα μπορούσαμε να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, για τη μικρή οργανισμοί προσφύγων πρωταγωνιστούν σε αυτό. Έχουμε σημαντικότητε εμπειρίε. Σε εμά υπάρχει το Μουσείο ε, Εξερεύνηση που δεν υπάρχει σε άλλε χώρε και παρουσιάζει σε παιδιά ε, νέα της ιστορίας των προσφύγων με τρόπο καλλιτεχνικό. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε όλα αυτά, να ενισχύσουμε τα δίκτυα προσφύγων καλλιτεχνών, ε, εκπροσώπων ε, του πολιτισμού, συγγραφείς για παράδειγμα. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, να τους εντάξουμε στο ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου θα εξετάσουμε, θα δούμε όλοι στους διαφορετικούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και πρέπει να δούμε και αυτούς τους ανθρώπους με αυτή τη νέα ιδιότητα. Ευχαριστώ, χαίρομαι για αυτή την ακρόαση. Ήταν πολύ καλή πρωτοβουλία, διότι ο πολιτισμός σημαντικός για τους μετανάστες, εντάξει μεταναστών, μειονοτήτων ε, και για μια ειρηνική κοινωνία. Χρειαζόμαστε ειρήνη και αλληλεγγύη, κάτι που λείπει. Πρέπει να το προωθήσουμε αυτό. Χάρη στην υπέροχη ε, κυρία που ταγούδησε πριν, ε, ε, ε, αισθανθήκαμε τι ήθελε να πει και θέλαμε να χορέψουμε και όλα με το τραγούδι της. Και η Χάρμα Άρμα χαίρομαι που αναφέρθηκε, ήταν, είναι φιλόσοφος γυναίκα και πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνει κανείς να ενεργοποιηθεί, αν είναι κανείς στη μειονότητα ή παρείας, ε, τι αντίκτυπο έχει αυτό για την κοινωνία και για τις μειονότητες. Να δραστηριοποιείται κάποιος και πάντα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Είμαι λευκή, Γεννήθηκα στη Δυτική Ευρώπη, έχω καλή εκπαίδευση, δεν είμαι φτωχή, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι που υποφέρουν, που είναι φτωχοί και κυρίως οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πολλά προβλήματα. Το ξέρουμε την κατάλληλη εκστατεία ότι είναι δύσκολα τα πράγματα όταν είναι κανεί στη θέση που είμαι εδώ. Υπάρχουν προβλήματα στι ευρωπαϊκές κοινωνίες και στον κόσμο. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Λιβύη, στο φτυχτό καθεστώ του Ασάτη, λέει ο Τραμπ. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά ε, την παρενόχληση, ε, την έμφυλη παρενόχληση κλπ. Λοιπόν, και στην ευρωπαϊκή κοινωνία, και σε όλα τα κράτη-μέλη επίση, και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν τα προβλήματα. Άρα είναι το ερώτημα πώ να βρούμε μια καλή λύση για του πρόσφυγε και του μετανάστε. Και είμαι πεπισμένη ότι χρειαζόμαστε πολιτικό άσυλο για του πρόσφυγε και νόμους μεταναστεύσεως με ποσοστώσεις για ε, τους ε, νόμιμους μετανάστες που έρχονται εδώ για εργασία. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους ε, ψηφοφόρους γι' αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που προωθούν οι ακροδεξοί στη Γερμανία για τους μετανάστες. Αυτό που είπατε αφορά τη δραστηριοποίηση και να αποκτήσει κανεί τη δύναμη, μόνο τότε μπορεί να είναι ενεργό πολίτη κανεί. Αλλιώ δεν τα καταφέρνει. Αν είναι απλώ θύμα, δεν μπορεί να δρά υπεύθυνα. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τα προβλήματα με διαφόρους ψηφίζουν ε, τους δεξιούς και λεπέν, τους άντρες, αλλά υπάρχουν και γυναίκες. Και σε κάποιο βαθμό είναι πρόβλημα με τους άντρες που ψηφίζουν ακροδεξιό. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτούς ανόητους άντρες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, καμιά φορά αποτελούν ένα τμήμα του προβλήματος. Μ' αρέσουν οι προτάσεις σας. Με το πρόγραμμα Εράσμος πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στα θέματα αυτά και να το χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα. Με καλύτερη πρικοδότηση ελπίζουμε το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Υποστηρίζω τις προτάσεις σας. Πολύ επικοδομητικές. Και ελπίζω σημερινή ακρόαση θα επηρεάσει ε, το Κοινοβούλιο και τις εργασίες του Κοινοβουλίου και την προσέγγισή μας. Ευχαριστώ. Αλλά επειδή δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο... Α, α, α θέλεις και εσύ. Μπόγκταν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, παρουσίαση που κάνατε της πολύ ενδιαφέρουσας ε, έρευνας. Αυτό που κάνουμε είναι να ασχολούμεθα με τα διάφορα προγράμματα, τα πολιτισμικά. Αναφερθήκατε στην πρόσβαση, στη χρηματοδότηση αυτών και κάνατε κάποιες συστάσεις. Ταυτόχρονα αναφερθήκατε σε νέες λύσεις και νέες πλατφόρμες δραστηριοποίησης για μένα είναι σημαντικότατη η ένταξη των προσφύγων, η επίδειξη αλληλεγγύης προς αυτούς. Θα πρέπει να δούμε ότι αυτοί που έρχονται εδώ είναι οι ίδιοι με μας. Όταν μιλάτε λοιπόν για νέα προγράμματα, δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες για να συμπεριλάβουμε και τον αθλητισμό που είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού. Γιατί το λέω αυτό, διότι με ενδιαφέρει πολύ αθλητισμός, καλύπτεται από το έρασμο συν, αφορά την φυσική δραστηριότητα. Για να πετύχουμε τους στόχους θα είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε και τον αθλητισμό. Με τον συνάδελφο τον κύριο Φίσας ξεκινήσαμε κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό θέλουμε να εντάξουμε κοινωνικά τους πρόσφυγες. Παρακολουθούμε την εφαρμογή ε, του όλου προγράμματος και για περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος θα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιείται ο αθλητισμός για την ένταξη των νέων ανθρώπων, να αποκτούν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση επίσης. Εδώ μεγάλος Χρειάζεται και γλωσσική εκπαίδευση όμως για να ξεφύγουν από κάποια εμπόδια για να μην εξωστρακίζονται και να μην στιγματίζονται. Τι κάνετε λοιπόν στον αφορά τον αθλητισμό είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ η Τζούλι Βόρτ για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η πρωινή παρουσίαση και ήμουν υπερήφανη που άκουσα τόσες βρετανικές φωνές που ε, ακολούθησαν μια πολύ ε, συναισθηματική προσέγγιση στον αφορά τους ε, πρόσφυγες. Έχω εργαστεί στο θέατρο και είχα συνεργαστεί με περιθωριοποιημένες κοινότητες και είναι υπέροχο να βλέπω το έργο που γίνεται στον τομέα των τεχνών και της δημιουργίας και τη δραστηριοποίηση τομείς αυτούς και να βλέπω εκπροσώπους εδώ, να το βλέπω να συμβαίνει. Τραγουδήσατε σε αυτό το χώρο, ήταν υπέροχο. Επίσης, ευχαριστώ που αναφερθήκατε στους Ουγγενώτους. Ήταν Ουγγενώτη η προγονή μου. Άρα το παρελθόν μου, το ιστορικό μου είναι από πρόσφυγες. Κανείς δεν χρειάζεται να πάει πολύ μακριά στην ιστορία του για να βρει ότι κάπου στους προγόνους τους υπάρχουν πρόσφυγες. Και οι Ουγγενώτοι ήταν διωγμένοι Γάλλοι που έπρεπε να φύγουν και έδωσαν τη λέξη, ε, ε, ενέταξαν τη λέξη πρόσφυγα στο λεξιλόγιο μας. Οι πρόγονοί μου κατέληξαν στο ε, Νότιγχαμ και έφεραν τα κεντητά στο Νότιγχαμ και υπάρχει ακόμα αγορά κεντημάτων στο Νότιγχαμ. Και ήταν βάση του πλούτου της πόλης. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό όταν μιλάμε για τις πρόσφυγες δεν έρχονται ξεφεύγοντας με τίποτα στα χέρια τους, έρχονται με εξαιρετικές ε, δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, φέρνουν μεγάλο πλούτο και δυνατότητες ε, στις κοινωνίες μας και στις ε, κοινότητές μας. Πριν από δέκα μέρες περίπου ήμουνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετείχα στο φεστιβάλ, σε ένα φεστιβάλ που ετοιμάζεται κάθε χρόνο. Ήμουν στο Νιου Κάσλ για να συμμετάσχω στην εκδήλωση να μάθω τους πρόσφυγες στην βορειοανατολική Αγγλία ποιες είναι οι παραδόσεις τους, παραδόσεις τους, ποιες ήταν οι φρικτές τους εμπειρίες και πώς αισθανόταν να βρίσκονται στη Βρετανία με το ρατσισμό που ξέσπασε μετά το δημοψήφισμα στη Βρετανία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που τονίσατε το ότι έχουν ευθύνη οι πολιτικοί όταν μιλάνε χρησιμοποιούν λόγια, λέξεις, εικόνες όταν δρούν και όταν δημιουργούν ε, αρνητικό περιβάλλον μέσω των νόμων που θεσπίζουν. Εγώ είμαι μέλος ε, του κινήματος του αντιρατσιστικού του ευρωπαϊκού και είμαι συνειδητία του Eli Wiesel, του δικτύου, που ευαισθητοποιεί ε, για θέματα γενοκτονίας και άρνησης γενοκτονίας. Και κάτι από αυτό που συμβαίνει στα βήματα προς τη γενοκτονία είναι η κατάρτιση καταλόγων ανθρώπων. Πρόσφατα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε δύο παραδείγματα. Άμπερ Ράντ πρότεινε ότι όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ετοιμάζουν καταλόγους ανθρώπων από άλλες χώρες, καταλόγους και πρόσφατα συντηρητικός βουλευτής, ο Chris Heaton Harris νομίζω, έγραψε σε όλους τους των Πανεπιστημίων ζητώντας καταλόγους ανθρώπων, ατόμων που ασχολούνται ε, με ευρωπαϊκές μελέτες, σε δίδασκαν ευρωπαϊκές μελέτες. Ξεκίνησαν με καταλόγους οι γενοκτονίες. Ε, και αυτό που κάνει ο Ερντογάν στην Τουρκία δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχαν κατάλογοι ανθρώπων που είναι ανεπιθύμητοι, Φερρυπίν, που κάνουν πράξεις που θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι απειλητικές πράξεις εναντίον τους. Ευχαριστώ που επιστήσατε την προσοχή στους επικίνδυνους καιρούς που περνάμε όταν οι δεξιοί πολιτικοί ε, δαιμονοποιούν ε, κάποιους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάθιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρει παρατηρήσει θέλω να κάνω. Μου επιτρέπετε να ευχαριστήσω ωστόσο την γραφή που ήρθε μαζί μα εδώ. Να σα συγχαρώ. Να συγχαρώ και την κυρία που τραγούδησε νωρίτερα. Το πρώτο που έχω να πω έχει να κάνει με το εύρος αυτών των εκθέσεων. Εργάζονται όλα αυτά τα έργα με ε, πρόσφυγες ε, και θα ήθελα αυτό να επεκταθεί και στους μετανάστες και οι μετανάστες έρχονται στις χώρες μας αντιμετωπίζοντας τα ίδια προβλήματα με τους πρόσφυγες ε, επίσης ε, έχουν ε, εξίσου πολλά να προσφέρουν από πολιτισμική άποψη, από άποψη καλλιτεχνικών ικανοτήτων, ως κοινότητες και ως άτομα. Θα ήθελα λοιπόν αυτές ε, οι πολύτιμες προσπάθειες να επεκταθούν όχι μόνο από τους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Το δεύτερο που θέλω να πω, φοβάμαι, δεν θα είναι τόσο επικοδομητικό. Οι πρόσφυγες ε, βρίσκονται σε μια τρομακτική κατάσταση, αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες ε, στις χώρες τους, τρομακτικές και το γνωρίζουμε όλοι ότι πολλοί από αυτούς δεν επιβιώνουν ως πρόσφυγες. Είναι συνεπώς απολύτως αναγκαίο η βοήθεια που τους προσφέρουμε να είναι η σωστή. Αν τους προσφέρουμε λάθος βοήθεια, μπορούμε να τους οδηγήσουμε σε επιδείνωση της κατάστασής τους. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε πολιτική θα πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία. Να συγχαρώ του ε, συντάξει τη τρίτη έκθεση για όλα τα δεδομένα που έχουν συμπεριλάβει και τι πληροφορίε. Βοηθά πολύ. Αλλά οι συντάκτε των πρώτων δύο εκθέσεων ε, δεν είναι ιδιαίτερα αξιέπαινοι. Εξίσου αξιέπαινοι. Μα έδωσαν πολλέ γνωμοδοτήσει, έκαναν διάφορε υποθέσει, χωρί όμω να βασίζονται αυτέ σε στοιχεία. Να σα δώσω δύο παραδείγματα μεταξύ πολλών. Στην πρώτη έκθεση, ε, όταν. Ε, μιλάμε για την ε, Αυστραλία. Γράφτηκε ότι κανένα πολιτισμικό έργο για τους πρόσφυγες που δεν συμπεριέλαβε τους πρόσφυγες ε, δεν εστιαζόταν στην ευημερία τους. Και στη δεύτερη έκθεση υπήρχε ένα σχόλιο ότι τα έργα επηρεάζονται από τη σιωπηρή και ιστορικά σωρευμένη γνώση μνημών από ρατσιστικέ και απεικιοκρατικέ ιδέες. Ναι, μπορεί να ισχύουν αυτές οι δηλώσει, μπορεί και όχι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τέτοιους ισχυρισμού. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας λέει ότι ένα έργο ε, χαρακτηρίζονταν από το ένα ή από το άλλο και ότι αυτό οδήγησε στην επιτυχία ή όχι του. Ε, τίποτα λοιπόν δεν στηρίζει τον ισχυρισμό ότι πολλοί άνθρωποι που εργάζονται με πρόσφυγες αισθάνονται έτσι. Όταν κάνουμε λάθος, σε τέτοιες περιπτώσεις υποφέρουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες. Αν με επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε να ολοκληρώσω με μια πολιτική δήλωση. Στην πρώτη έκθεση αναφερόταν και πάλι στην παρουσίαση ότι οι δεξιοί πολιτικοί έχουν κάνει τέτοια σχόλια. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι και οι αριστερές κυβερνήσεις έχουν ένα φρικιαστικό ιστορικό γενοκτονιών και εθνοκαθαρσεών. Το να λέμε λοιπόν τέτοια πράγματα είναι αντιπαραγωγικό διότι όσοι είναι λιγότερο ανεκτικοί από εμένα θα πούν ότι αυτά είναι αριστερολογίες και θα τα απορρίψουν. Ε, ε, ενώ έχουμε πολύ θυμολικό εδώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Vielen herzlichen Dank. Η Χέλγα. Θα αποτίσω φορή τιμή στη Χάνα Άρεν και τη συζήτηση με τον εξή τρόπο. Τον επόμενο χρόνο που θα είναι το έτος της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Επιτροπή μας ή οι γυναίκες συντονίστρες θα έπρεπε να κάνουμε μια κοινή συζήτηση με γυναίκες φιλοσόφους την Άγνα Σέλα και μια καθηγήτρια μαύρη από το Ρότερνταμ που ξέχασα το όνομά της η Νίλη Φέγγελ, η Κάρολ Νέγκε, Χέρτα Μιούλα και ίσως να υπάρξουν και κάποιες άλλες από την Αφρική ή από άλλες υπήρους. Θα πρότεινα το χρόνο είτε εμείς ως ε, γυναίκες ε, μέλη του Κοινοβουλίου είτε η Επιτροπή μα συνολικά μετά την ακρόαση αυτή νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε μια υψηλού επίπεδου ε, διάσκεψη με τις ε, ε, ευφιέστερες γυναίκες ε, που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε να επανέλθω στις εμπειρογνώμονές μας. Ε, με τη σειρά θα σας δώσω το λόγο και ο καθένας μπορεί να απαντήσει σε όποια από τα θέματα ετέθησαν θεωρεί ότι είναι καλό να το κάνει. Λοιπόν, σας παρακαλώ πέντε λεπτά περίπου η κάθε μία. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ε, προκλήσεις αν θέλετε και την υποστήριξη του έργου μας. Για τα στοιχεία πρώτον να απαντήσω. Έχει πολλές μορφές το στοιχείο. Καμιά φορά είναι δράση σε συμμετοχή. Δεν είναι πάντα αριθμός και κατάλογοι που μπορούν να μας αποδείξουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ίσως μπορεί να δείτε ότι ο Τζον Ντούι είπε ότι υπάρχει ένα μικρό φάσμα πραγμάτων που μπορεί να καλύψει η θετικιστική προσέγγιση. Θα πρέπει εδώ να έρθουμε και να σχορέψουμε, μας ενθαρρύνατε να το κάνουμε. Έρχομαι στον αθλητισμό. Ζωτικός τομέας η συμμετοχή όλου του σώματος. Όχι μόνο τις ομιλίες τη συζητήσεως, είναι ζωτική σημασία. Και ιδιαίτερα άμα σκεφτούμε ότι θέλουμε την ευημερία ω κοινωνία. Ο αθλητισμός κάνει καλό σε όλου. Όσο πιο πολύ θα μαζί, τόσο το καλύτερο. Τα τελευταία δέκα χρόνια στις εργασίες μου στο πολιτιστικό, το τομέα μου πρόσφυγε θέατρο, χωρό κλπ. Είδα ότι βελτιώθηκε μέσω της συμμετοχής και η λειτουργία της καρδιάς μου και η πίεση μου. Σας το συστήνω ένθερμα. Λοιπόν, θα πρέπει ο πολιτισμός να θεωρηθεί σαν αθλητισμός. Είναι πάρα πολύ καλό εγχείρημα αθλητισμός. Τον Άντι Μάρι και τον Ρότζο Φέντερερ να τους βλέπετε να παίζουν τένις για να, να δείτε λοιπόν τη γεωμετρία εν κινήσει. Ευχαριστώ που σημειώσατε αυτό που είπαμε για τη γλώσσα. Είναι κρίσιμη η σημασία της. Πάντα περνάει από σημειολογικές αλλαγές. Είδαμε από την κρίση του 2015 που είχαμε αρκετέ χώρε για υποδοχή των προσφύγων και πολλοί πνίγηκαν στην Μεσόγειο. Η γλώσσα, η διατύπωση που χρησιμοποιείται ε, ήταν αρκετά ανησυχητική και εξακολουθεί να είναι ανησυχητικό το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται. Αλλά άλλαξε σημειολογικά η έκφραση και στη χώρα μου σίγουρα. Έγινε αποδεκτό να μιλά κανείς για μετανάστες και χρησιμοποιείται και η λέξη πρόσφυγε στη Σκοτία, στη χώρα μου, οι πρόσφυγες και η ομάδα μας είναι οι νέοι Σκοτσέζοι. Αυτό προτιμούν να χρησιμοποιείτε. Πρέπει να προσέχουμε τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για νέους Ευρωπαίους. Τι θα σήμαινε να χρησιμοποιούμε τη λέξη νέοι Ευρωπαίοι, τις λέξεις νέοι Ευρωπαίοι. Υπέροχα τα σχόλια που ακούστηκαν. Αναφέρθηκαν στο από πού ε, προέρχεται κανείς και τι γίνεται στην Ιταλία. Είναι σημαντικά θέματα, αλλά δεν είναι η πρωτή της σημασίας. Στο έργο μου δεν ρωτάω σε κάποιον, δεν ζητάω από κάποιον να μου πει το ιστορικό του. Το κάνουν οι γραφειοκράτες και οι δικηγόροι. Εκεί στο νομικό πλαίσιο χρειάζεται αυτό. Αν θέλουμε να κατασκευάσουμε μια οικονομία που μοιραζόμαστε ιστορίες, δεν πρέπει να παρουσιάζουμε καλές ή κακές ιστορίες ενό ταξιδιού μόνο να λέμε περισσότερα. Άρα, τι μπορεί να παίξει κανείς, μουσικό όργανο, ε, κάποιο, κα, ασχολείται με κάποιο σπορ. Ε, μπορείτε να θέλετε να μου πείτε, αυτό είναι υπέροχο που φοράτε, ε, πείτε μου την ιστορία που το πήρατε κλπ. κλπ. Πρέπει να λέμε άλλες ιστορίες, είναι το πνεύμα. Ευχαριστώ κύριο Νέντερμαϊα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα σχόλιά σας για τις γυναίκες φιλοσόφους. Θαυμάσιο θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια εκδήλωση. Θα έπρεπε να είναι πολυτομιακή προσέγγιση, να αντιμετωπίσουμε, να συμπεριληφθούν άτομα ε, που υφίστανται διακρίσεις όχι μόνο για λόγους φίλου, αλλά και ε, σεξουαλικής ταυτότητας και εθνικότητας, οτιδήποτε περιθωριοποιεί τους ανθρώπους. Αυτά που είπατε για την ε, έμεση γνώση σε σχέση με το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα έπρεπε η Ευρώπη να ξαναδεί την ε, ιστορία, την επικοκρατία, το ρατσισμό, την ιστορία της. Γιατί δεν έχουν εξαφανιστεί. Εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν πολλές μελέτες μεταπικιακές που το αποδεικνύουν. Ο βραβευμένος με το Νόμπελ Οικονομίας φέτος ακριβώς ασχολείται με τα θέματα έμεσης και ασυνείδητης γνώσης που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας. Το θέμα για τον αθλητισμό. Θα έπρεπε να συνδυάσουμε τα προγράμματα για τον αθλητισμό με την εκπαίδευση. Μια πολυτεμιακή προσέγγιση είναι αναγκαία. Οι πρόσφυγες είναι ανθρώπινα όντα και θέλουν να ε, έχουν καλό επίπεδο ζωής. Και για να έχεις ε, καλό επίπεδο ζωής πρέπει να ε, ασχολείσαι με πολλά πράγματα. Δεν αρκεί μόνο ο πολιτισμός. Κάτι άλλο. Και αυτό που είπε και η κυρία από την Ιταλία. Βεβαίως πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Γιατί ναι, μπορεί να έχει περάσει κρίση, ή τουλάχιστον ελπίζουμε. Αλλά όσοι έχουν έρθει στην Ευρώπη δεν πρέπει να είναι απλώς σε επισφαλή κατάσταση. Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για ε, κοινωνική άνοδο, να μπορέσουν οι πρόσφυγες να επιτύχουν πράγματα στη ζωή τους και να σταματήσουμε να μιλάμε για ένταξη γιατί η ένταξη στην ουσία περιθωροποιεί τους πρόσφυγες. Δηλαδή, το να μιλάμε για ένταξη. Σε πόσες χώρες υπάρχουν τέτοια προγράμματα, με ρωτήσατε. Βεβαίως, ε, κυρίως η Γερμανία και η Σουηδία και άλλες χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, που είναι οι κύριες χώρες υποδοχής προσφύγων, εδώ υπάρχει η περισσότερη πυκνότητα τέτοιων προγραμμάτων, δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες, που χρηματοδοτούνται από διάφορους ε, φορείς. Ελπίζουμε και ο ιδιωτικό τομέα να χρηματοδοτήσει. Ενώ σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν πολύ λιγότερα τέτοια προγράμματα. ετέθη το θέμα ότι οι πρόσφυγες έχουν διαφορετικές ε, προελεύσεις. Αυτό βέβαια δημιουργεί προβλήματα για την απονομή του καθεστώτος ε, πρόσφυγα σε κάποιον. Αλλά ξέρετε, οι περισσότεροι που έρχονται στην Ευρώπη έρχονται για τους ίδιους λόγους, οπότε το θέμα είναι λεπτό. Πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούις ή η κυρία Μάρτιν. Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ανέφερε ο κ. Μάθιος όταν μίλησε για τη σωστή βοήθεια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γίνεται πολλή δουλειά, πολλές προσπάθειες. Κατά την προσωπική μου άποψη όμως, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα για να ακούσουμε τις απόψεις, ε, τις φωνές των μεταναστών, να καταλάβουμε τι ακριβώς χρειάζονται, γιατί όλοι θεωρούμε δεδομένο ότι θέλουν να ενταχθούν και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ορισμένοι δεν το επιθυμούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό επιχείρημα σε αυτή τη συζήτηση και εντό των έργων τα οποία χρηματοδοτούνται και οργανώνονται στι ερευνέ μας ε, ανακαλύπτουμε ότι αυτή η πτυχή πολλέ φορέ ε, αγνοείται ή παραβλέπεται. Ε, οπότε είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου για την αλληλεγγύη που βλέπουμε εδώ στην αίθουσα από ευρωβουλευτές διαφόρων ε, χώρων και βλέπω ότι όλοι κατανοούν το ζήτημα με τον ίδιο τρόπο και νιώθω ότι υπάρχει ένα κοινό όραμα για το τι χρειαζόμαστε. Ε, χαίρομαι λοιπόν που το βλέπω αυτό. Για τον αθλητισμό σίγουρα, ναι ξέρετε ο πολιτισμός έχει κεφαλαίο που ε, περιλαμβάνει ένα σωρό όλους τους τομείς, είναι πολύ σημαντικός. Ο πολιτισμός περιλαμβάνει και τον αθλητισμό και ένα σωρό άλλα πράγματα και είναι σημαντικό να ηγείται αυτής ε, ε, ο κόσμος, οι κοινότητες ε, και να συμπεριλαμβάνεται και ο αθλητισμός. Τώρα για τα στοιχεία που αναφέρατε, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ως βάση από τα στοιχεία, αλλά και στοιχεία που να δείχνουν τα αποτελέσματα. Και αυτό είναι το δύσκολο, διότι απαιτείται κάποιο πλαίσιο ευέλικτο αρκετά ώστε να μπορούμε να δείξουμε όχι μόνο τα αποτελέσματα των προϊόντων ε, στους ενδιαφερομένους αλλά και τις διαδικασίες ε, το ταξίδι που έκαναν όσοι συμμετείχαν ε, τι έζησαν οι συμμετέχοντες σε όλα αυτά τα προγράμματα οι εμπειρίες αυτές είναι το κλειδί ευχαριστούμε κυρία Κώστα για τα σχόλιά σας για το πρόγραμμα αυτό από την ενδιάμεσα ε, αναθεώρηση του Creative Europe του Erasmus Plus ε, ε, μαθαίνουμε πορίσματα των ερευνών Πρέπει, όπως βλέπουμε, ε, να ρωτάμε τους, μετα... τους πρόσφυγες ε, τι μπορείτε να κάνετε, τι θέλετε να γίνει. Αυτό θα συμπεριλάβουμε στα νέα γενιά προγραμμάτων ερωτήσεις τέτοιες. Και τέλος, ε, για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπάρχει ένα κομμάτι στην έκθεσή μας για αυτό το θέμα. Αποτελεί ευκαιρία να μιλήσουμε για την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά ως ανθρώπινα όντα παγκοσμίω ε, είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν του πάντε. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το ζήτημα, είναι παγκόσμιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμότατα όλες τις, όλους τους εμπειρογνώμονές μας και εσάς ε, κυρία μου για την ε, μουσική σας συμβολή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν με τόσο ενδιαφέρον και έκαναν τόσες προτάσεις που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω εργασία μας. Φυσικά θα συζητήσουμε τώρα τα επόμενα βήματά μας. Την πρόταση της Χέλγα θα τη συζητήσουμε με τους συντονιστές για να δούμε τι θα μπορούσαμε να Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία όλων σας. Ευχαριστώ που συμμετείχατε στη συζήτηση και άλλη μια φορά. Ευχαριστώ και το τμήμα πολιτικής που οργάνωσε και προετοίμασε αυτή την ακρόαση. Νομίζω ότι ήταν ε, ιδιαίτερα θετική. Όλοι μάθαμε. Ευχαριστώ πολύ.